Dear colleagues, probably is time to... Αγαπητοί συνάδελφοι, ήρθε η ώρα να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Και θα αρχίσω αμέσως με το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται χωρίς τροποποίησης. Έχω να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις στο σημείο 2. Πρώτον, θα οργανώσω θα οργανώσουμε μια εκτακτή συνεδρίαση στο Στρασβούργο τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στις 7 για να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς, ο οποίος είναι υπεύθυνο για την ε, εφόρο ανάπτυξη. Σήμερα έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες και ως ήθιστε ηλεκτρονικά μεταδίδεται η συνεδρίασή μας μέσω του διαδικτύου τώρα περνάμε στο κυρίω σημείο στην ημερήσια διαταξή μας, που είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον Μάρος Σεύκοβιτς. Είναι υπεύθυνο για την Ενεργειακή Ένωση, για το προσεχές στρατηγικό πλαίσιο για την Ενεργειακή Ένωση. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Αντιπρόεδρο Σεφκοβιτς. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Επιτροπή μας από τότε που ανέλαβε την Αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως υπεύθυνο για την Ενεργειακή Ένωση. Στις 20 Φεβρουαρίου 25 Φεβρουαρίου του 2014 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το πλαίσιο για την ενέργεια και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια πλήρως λειτουργούσα και συνδεδεμένη αγορά ενέργειας προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση ενεργειακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προτεραιότητες αυτές αντικατοπτρίζονται στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015 και με τη σημερινή μας ανταλλαγή απόψεων θα επικεντρωθούμε στις προτεραιότητες, ιδιαίτερα αριθμό 3 που αναφέρεται στην αντοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις ενεργειακές προκλήσεις βάσει των όσων εγκρίθηκαν στις 25 Φεβρουαρίου. Το στρατηγικό πλαίσιο θα επικεντρωθεί στην ε, ενεργειακή ασφάλεια, στις αγορές, στην απόδοση ενέργειας, την αποτελεσματικότητα του ενεργειακού μείγματος και προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πρώτη στον κόσμο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα με τον Αντιπρόεδρο. Ισοτική σημασία επίση, όταν εξετάσουμε τι κλιματικέ αλλαγέ, είναι το σχέδιο τη Επιτροπή για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και το ETS και τα σχετικά προγράμματα για την, ε, τους πληστηριασμούς εκπομπών διοξίδιου του άνθρακα. Και όλα αυτά προετοιμάζοντας τη διάσκεψη για το κλίμα στο Παρίσι. Έπειτα μας ενδιαφέρει η σύνδεση με μια αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική. Ξέρετε ότι η Επιτροπή μας ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τις αρνητικές συνέπειες από την ρήπανση και πιστεύει ότι πρέπει να προωθήσουμε νομοθεσία για να αποφύγουμε τους ρηπαντές. Θέλουμε να συνεχίσουμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάλληλη νομοθεσία που να είναι δεσμευτική στα πλαίσια του τις δράσεις του 7ου προγράμματος πλαισίου, που είναι μεγάλη προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θέλουμε επίσης να μάθουμε περισσότερα για τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοινώθηκαν ήδη στα πλαίσια του προγράμματος εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015 όσον αφορά τους ατμοσφαιρικούς ρηπαντές. Και αυτό για να δούμε τι νομοθετικά μέτρα θα ακολουθήσουν. Προσβλέπουμε σε ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα αυτά τα θέματα και δίνω το λόγο στον Αντιπρόεδρο ευθύ αμέσω για τι εισαγωγικέ του παρατηρήσεις. Ε, Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Νορβηγικού Κοινοβουλίου που είναι εδώ σήμερα. Τους ευχαριστώ όλους που ήρθαν να επισκεφθούν την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λαβία, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές ε, και φίλοι από την Ορβηγία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευγενή σας πρόσκληση να παρευρεθώ σήμερα εδώ και να έχω τη δυνατότητα να παρακολουθήσω την έκτακτη αυτή συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΝΒΗ. Διότι θα μου επιτρέψει να μοιραστώ μαζί σας κάποιους συλλογισμούς σχετικά με το πώς ετοιμάζουμε και οριστικοποιούμε το πλαίσιο που θέλουμε να σας παρουσιάσουμε μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου. Εκτιμώ λοιπόν το ενδιαφέρον σας για την Ενεργειακή Ένωση. Χθες είχα την ευκαιρία να έχω μια παρόμοια ανταλλαγή απόψεων με τους συναδέλφους σας από την Επιτροπή Ήτρε. Ήταν πολύ χρήσιμη η συνάντηση αυτή. Δεν έρχομαι μόνο να σας παρουσιάσω τις ιδέες μας, έρχομαι να ακούσω και τις δικές σας ιδέες, τις ανησυχίες σας σχετικά με τις κύριες προτεραιότητες της Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη. Πιστεύω λοιπόν ότι έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και καλή συζήτηση. Η Ενεργειακή Ένωση θεωρείται μια από τις κύριες προτεραιότητες της νέας Επιτροπής Juncker και γι' αυτό χαίρομαι που μπορούμε σήμερα να έχουμε αυτή τη συνάντηση. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Μας απομένουν κάποιες εβδομάδες μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου, την ημερομηνία που σκοπεύουμε να υιοθετήσουμε το πακέτο για την Ενεργειακή Ένωση. Ξέρω ότι κάποιοι από εσά εκπονείτε γραπτές συνεισφορές και προσλέπουμε στην παραλαβή του από εσά. Ε, προσλέπουμε όμως και στις προσωπικές διαβουλεύσεις τις ε, προφορικές σας παρατηρήσεις σήμερα, αλλά και στην συνέχεια της διαδικασίας διαβούλευσης που θα έχουμε με κάποιους από εσά και που θα πραγματοποιηθεί και στη ρίγα. Αξιότιμοι βουλευτές, αγαπητοί φίλοι, όταν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε τις προτάσεις του για την αλλαγή του τρόπου εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι πρέπει να γίνουμε μεγαλύτεροι στα μεγάλα θέματα, να κάνουμε περισσότερα δηλαδή για τα σημαντικά θέματα. Και αναφέρεται στις πολιτικές που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ζωές των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι θέλουμε να διασφαλίσουμε καλές τιμές θέρμανσης. Πρέπει όλοι ε, να έχουν πρόσβαση στη θέρμανση και να έχουμε σταθερότητα στις τιμές. Ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε οι εταιρείε μας συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να μπορούν να αγοράζουν ενέργεια με ανταγωνιστικές τιμές και να γίνουν η πραγματική μηχανή ανάπτυξης και να δημιουργήσουν τις θέσεις εργασίας που ε, θα χρειαστούμε στο μέλλον. Θέλουμε όμως και ο καθένας από το και από το Πόρτο, να μπορέσει να εφαρμόσει επιτυχώς ε, λαμπρές ιδέες στην Ευρώπη και να μην χρειάζεται να πάει στις ΗΠΑ ή στην Κίνα. Θέλουμε η Ευρώπη να παραμείνει επικεφαλής στον τομέα αυτόν. Θέλω όμως επίσης να διασφαλίσω για τα ε, εγγόνια μου στην Πρατισλάβα, για τα παιδιά σας ε, στην Ευρώπη, στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες. Θέλουμε λοιπόν να φροντίσουμε τα παιδιά αυτά να μην χρειαστεί ποτέ να πληρώσουν το τίμημα για τα περιβαλλοντικά λάθη των προηγούμενων γενναίων. Αυτοί οι στόχοι μπορεί να φαίνονται πολύ φιλόδοξοι, είναι όμως εφικτοί και πιστεύω ότι τώρα υπάρχει το πολιτικό κλίμα για να θέσουμε σε κίνηση την Ενεργειακή Ένωση. Η παρούσα γεωπολιτική κατάσταση, στην οποία σίγουρα θα αναφερθούμε στη συζήτησή μας, ε, θα αναφερθούμε ιδιαίτερα στα ανατολικά μας σύνορα. Η κατάσταση αυτή λοιπόν ε, έχει θέσει την ενεργειακή ασφάλεια ακόμα πιο ψηλά στο θεματολόγιο της Ευρώπης η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ε, κλιματικό και ενεργειακό πλαίσιο για το 2030 έχει ανοίξει την πόρτα για μια φιλόδοξη συμφωνία στο Παρίσι και θα πρέπει να συζητήσουμε πώς μπορούμε να πετύχουμε καλά αποτελέσματα στο Παρίσι και να εφαρμόσουμε με αναλάβει στο πλαίσιο ε, του προγράμματος Ευρώπη 2020. Οι συζητήσεις στη Λίμα ήταν πολύ δύσκολες, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπόρεσε να μιλήσει με μία φωνή. Είμαστε λοιπόν φιλόδοξοι ότι θα μπορέσουμε στο Παρίσι να πετύχουμε μια καλή συμφωνία. Και βέβαια έχουμε τώρα μια νέα επιτροπή η οποία θα ε, ε, συνεχίσει να επιμένει στις προσπάθειες για μια ανθεκτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα επενδύσεων του Juncker ε, σκοπό έχει να ξεκλειδώσει τους ε, οικονομικούς πόρους για τον ενεργειακό τομέα και για νέα περιβαλλοντικά προγράμματα. Και νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ε, το νέο κλίμα στο οποίο βρισκόμαστε, δείχνουν και την αποφασιστικότητα της Κομισιόν για να πετύχουμε τους στόχους μας. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε τώρα επιτέλους μια πραγματική ευκαιρία να επιφέρουμε αλλαγές και να κάνουμε άλματα πρόοδου. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε για να δράξουμε αυτή την ευκαιρία. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να είμαστε και ειλικρινεί στη συζήτηση αυτή. Η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια Παρά την σημαντική πρόοδο, οι παρούσες ενεργειακές πολιτικές μας ε, δεν είναι βιώσιμες. Οι τιμές είναι πολύ ασταθείς και ε, έτσι οδηγούν σε ε, φαινόμενα κερδοσκοπίας βαχυπρόθεσμα και μη προβλεψιμότητα, αβεβαιότητα πιο μακροπρόθεσμα. Το μεγαλύτερο μέρος τη ενέργεια Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από χώρες που χρησιμοποιούν την ενεργειακή παροχή ως ε, πολιτικό μέσο. Μπορείτε να δείτε στι οθόνε πόσο εξαρτώμαστε από τις εισαγωγέ και πώς η εξάρτησή μας έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, θα πρέπει να είμαστε και ειλικρινεί και να αναγνωρίσουμε το γεγονό ότι είναι κατακαιρματισμένο το ενεργειακό μας σύστημα. Έχουμε 28 ξεχωριστά συστήματα και κάποια μέρη της Ευρωπαϊκής Υπήρου δεν έχουν ενταχθεί επαρκώς στο ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης. Στην οθόνη αυτή βλέπετε πόσες διαφορετικές πολιτικές έχουμε όσον αφορά τους μηχανισμούς δυναμικού στην Ευρώπη, τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ τους, αλλά και τι διαφορετικές προσεγγίσεις έχουμε. Και βέβαια όλα αυτά μας ε, στοιχίζουν πολλά χρήματα, ε, πολλά στοιχεία παρουσιάζονται. Το Παγκόσμιο Ευρωπαϊκό Φόρουμ ε, παρουσίασε βέβαια αμφισβητούμενα στοιχεία. αλλά είπε ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε 140 δισεκατομμύρια ευρώ εάν επικεντρωθούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακόμα και αν είναι αμφισβητήσιμα τα στοιχεία αυτά, θα έπρεπε να μας κάνουν να σκεφτούμε πώς μπορούμε να μεταρρυθμίσουμε τις αγορές μας. Ε, διότι έτσι θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και ε, να κερδίσουμε σε αξία. Επίσης, απόψε όταν θα γυρίσουμε στα σπίτια μας, οι περισσότεροι από εμά. Περιμένουμε να γυρίσουμε σε ένα σπίτι όπου όλα λειτουργούν. Σε ένα θερμενόμενο σπίτι με ζεστό νερό. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι, διότι αν ξανακοιτάξετε τη διαφάνεια θα, θα δείτε ότι το 10% των ε, νοικοκυριών μας ε, δεν ε, είναι φτωχά σε ενέργεια, δηλαδή δεν μπορούν να πληρώσουν το, τους λογαριασμούς και αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες διότι δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν κάτι το οποίο πριν λίγο καιρό είχαν και δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τις οποίες θα έπρεπε να μπορεί να καλύψει οποιοδήποτε νοικοκυριό. Το θέμα όμως εδώ πέρα δεν είναι μόνο οι καταναλωτές, ε, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και οι επιχειρήσει αντιμετωπίζουν τιμές ενέργεια σε φυσικό αερίου τριπλάσιες τη Αμερικής. Και αυτό είναι σημαντικό άκτος για τη βιομηχανία και την οικονομία μας. Και από τις 10 κορυφαίες εταιρείε ηλιακή ενέργειας στον κόσμο, καμία από αυτές δεν είναι ευρωπαϊκή. Έχουμε μείνει πίσω όσον αφορά την ανάπτυξη μπαταριών και αποθήκευσης ενέργειας. Η πρόοδος όμως σε αυτόν τον τομέα αποτελεί προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητά μας. Θα πρέπει λοιπόν ε, να προωθήσουμε τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας ε, στις μεταφορές ε, κλπ. Πρέπει όμως επίσης να είμαστε ειλικρινεί όσον αφορά την μεγάλη σπατάλη ενέργειας. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να οικοδομήσουμε την οικονομία χαμηλής, χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που θέλουμε και είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσά εδώ στην Επιτροπή ΕΝΒΙ τα γνωρίζετε αυτά. Όπως ε, σας είπα κατά τη διάρκεια της ακρόασής μου, εκπονούμε ένα πρόγραμμα ενεργειακής ένωσης όπου προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις τις οποίες ανέφερα. Και θα ήθελα αυτή η ενεργειακή ένωση να βασιστεί σε πέντε διαστάσεις. Μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου θέλουμε να προτείνουμε συγκεκριμένες ε, προτάσεις για κάθε ε, έναν από αυτούς τους τομείς. Ε, θα πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε την ενεργειακή ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας στην Ευρώπη. Πάνω από 400 δισεκατομμύρια το χρόνο αξίζει η, η ενέργεια που εισάγει κάθε χρόνο και θα πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές και να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις εγχώριες ε, πηγές ενέργειας. Επίσης θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ποικιλία όσον αφορά τις πηγές και τους προμηθευτές ενέργειας. Η ιστορία του νότιου διαδρόμου θα πρέπει να αποτελέσει και μάθημα και ευκαιρία. Ας, ε, λοιπόν, ας έχουμε λοιπόν περισσότερη διαφάνεια στις ε, συμβάσεις για το φυσικό αέριο και μαζί με την κυρία Μογκερίνη ας έχουμε καλύτερη ενεργειακή διπλωματία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δεύτερη διάσταση επικεντρώνεται στην οικοδόμηση μιας ενιαίας εσωτερικής ενεργειακής αγοράς η οποία να είναι ε, ανταγωνιστική. Χρειαζόμαστε ελεύθερη ροή της ενέργειας. Μια ενεργειακή αγορά όπου επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται παρέχοντας τις καλύτερες ε, τιμές για την ενέργεια με σωστές ε, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ε, πρακτικές. Και για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να εξελίξουμε τα εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό δεν θα γίνει εν μία νυχτή. Καταρχάς θα πρέπει να έχουμε ισχυρότερη περιφερειακή συνεργασία εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου με βάση κάποιες ε, ανταλλαγές απόψεων που είχα πρόσφατα με δημάρχους ε, και ενεργειακές εταιρείες. Ε, είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε την Ενεργειακή Ένωση μόνο με ενεργό συμμετοχή των πολιτών, των διαφόρων φορέων και των πόλεων. Θέλουμε ευφυείς πόλεις θα πρέπει να συμμετάσχουν οι πολίτες στη διαδικασία αυτή. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή τους ε, καθώς ε, και την ε, οικειοποίηση του προγράμματος από αυτούς. Η τρίτη διάσταση έχει να κάνει με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η καθαρή ενέργεια είναι αυτή που δεν έχει καταναλωθεί. Δηλαδή, λιγότερη κατανάλωση σημαίνει λιγότερη ρήπανση, λιγότερες δαπάνες και διατήρηση των ενεργειακών πηγών μας. Η βελτίωση την ε, ενεργειακή απόδοση ε, ε, ωφελεί τον, την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα καθώς και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το θέμα αυτό συνδέεται με τα κτίρια, με τις μεταφορές, με τα προϊόντα, την καθημερινή ζωή των πολιτών μας δηλαδή. Και αποτελεί σημαντική καινοτομία, αποτελεί όμως και σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας μια εντύπωση που μου δόθηκε κατά τις συναντήσεις των τελευταίων ημερών. Μου εξήγησαν ότι το 90% των κατοικιών μας ε, δεν είναι ενεργειακά αποδοτικό. Στην δεύτερη συνάντηση κάποιοι ιδιωτικοί επενδυτές ε, μου είπαν ότι θέλουν να επενδύσουν 9 ε, εκατομμύρια δολάρια ε, ε, σε νέα προγράμματα οικοδόμησης κατοικιών. Έχουμε λοιπόν ζήτηση, έχουμε και επενδυτές και θα πρέπει να συνδέσουμε αυτούς τους δύο παράγοντες μεταξύ τους ώστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διευκολύνουμε την διαδικασία που πιστεύω ότι θα μπορέσει να οδηγήσει σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρώπη. Η τέταρτη διάσταση συνδέεται με τη μείωση της ρήπανσης και την απαλλαγή από τους ανθρακούχες εκπομπές. Βρισκόμαστε καθοδόν προς το Παρίσι και η οδός αυτή οδηγεί και προς την Ενεργειακή Ένωση. Τον Οκτώβριο συμφωνήσαμε να μειώσουμε τις ε, εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% και αυτό δημιούργησε μια δυναμική ε, και στην Λίμα ο συναδελφός μου Άριος Κανιέτε μάλλον στη Λίμα ο συνεργάτης μου φρόντισε να μιλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση με μία φωνή και έτσι καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα τα οποία ανοίγουν το δρόμο για μια καλή συμφωνία στο Παρίσι. Η διπλωματία όμως είναι μία πτυχή, αλλά πρέπει και εμείς να εργαστούμε εδώ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους να πετύχουν καλή συμφωνία πάνω στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς ώστε οι εργασίες να μπορέσουν να συνεχίσουν πάνω στην αναθεώρηση του συστήματος εμπορία εκπομπών. Γνωρίζω ότι μας πιέζει ο χρόνος, ξέρω ότι καταβάλλετε σημαντικές προσπάθειες για να πετύχουμε καλά αποτελέσματα, αλλά όσο πιο σύντομα συμφωνήσουμε πάνω στο αποθεματικό για τη σταθερότητα τη αγορά, τόσο πιο σύντομα θα έχουμε τι προτάσει για την μεταρρύθμιση του συστήματο εμπορία εκπομπών και αυτό θα αποτελέσει πολύ σημαντικό επιχείρημα απέναντι σε όλου του εταίρου μα στι διαπραγματεύσει για μια καλή συμφωνία στο Παρίσι. Όπως είπε ο πρόεδρος Ιούνκερ, η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να είναι κορυφαία στον κόσμο όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας να απαλλάξουμε από ανθρακούχες εκπομπές τον τομέα των μεταφορών, που είναι ένα τομέα με όλο και αυξανόμενο μερίδιο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με την πέμπτη διάσταση, που συνδέεται με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία. Απαιτούνται τέτοιες επενδύσεις ε, όχι μόνο όσον αφορά τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας αλλά και για την μείωση των, της κατανάλωσης ενέργειας. Η τεχνολογική αιχμή στον τομέα αυτών θα δημιουργήσει τεράστιες ευκαιρίες εξαγωγών και έτσι θα έχουμε περισσότερες ε, θέσεις εργασίας και περισσότερη ανάπτυξη. Αξιότιμοι βουλευτές, αυτές είναι οι πέντε διαστάσεις μιας ολιστικής προσέγγισης που θέλουμε να έχουμε, που να καλύπτει πολλούς τομείς, όπως είναι οι μεταφορές, ε, το περιβάλλον, η ανταγωνιστικότητα, η γεωργία και η βιομηχανική πολιτική. Και δεν ασχολούμαι μόνο ε, εγώ με το θέμα αυτό. Έχουμε 16 γενικές διευθύνσεις και πολλούς επιτρόπους που συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία. Στο τέλος λοιπόν του Φεβρουαρίου θα δείτε το αποτέλεσμα μιας σημαντικής συλλογικής προσπάθειας, διατομιακής προσπάθειας. Θα ε, λάβετε λοιπόν προτάσεις από διάφορους τομείς. Οι προτάσεις αυτές θα αντιπροσωπεύουν ε, την ε, συλλογική προσπάθεια των επιτρόπων. Στο περιορισμένο χρονικό διάστημα που έχω στη διάθεσή μας. Δεν θέλω να ε, σας κουράσω με πολλές λεπτομέρειες, διότι νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια καλή συζήτηση και να δημιουργήσουμε τον κατάλληλο χώρο και να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας. Ξέρω όμως ότι ένα θέμα σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να κλείσω με το θέμα της διακυβέρνησης. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η Ενεργειακή Ένωση απαιτεί ισχυρό και αξιόπιστο σύστημα διακυβέρνησης. Πολύ προσεκτικά διάβασα την επιστολή που κάποιοι από εσά στείλατε προς τον Πρόεδρο Γιούνκερ, τον ε, Επίτροπο Άρια Κανιέτε και εμένα. Πολύ συχνά είχα βρεθεί στο Κοινοβούλιο και συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι το Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης θα πρέπει να παίξει ρόλο κλειδί την ε, εφαρμογή της Ενεργειακής Ένωσης. Ε, γι' αυτό σας υπόσχομαι ήδη τώρα ότι με την υιοθέτηση της ε, στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση από το Σώμα των Επιτρόπων η πρώτη μου κίνηση θα είναι να έρθω εδώ στο Κοινοβούλιο και να σας παρουσιάσω την ε, στρατηγική πλαίσιο και όχι μόνο θα σας παρουσιάσω τη στρατηγική αυτή, αλλά θα ζητήσω και την υποστήριξή σας, την οικειοποίηση αυτού του προγράμματος, γιατί είμαι πεπισμένος ότι μόνο με τη δική σας υποστήριξη θα μπορέσουμε να ε, εφαρμόσουμε στην πραγματικότητα την Ενεργειακή Ένωση και να έχουμε τα θετικά και συγκεκριμένα αποτελέσματα που θέλουμε για τους πολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτή την εισαγωγική παρουσίαση της καταστάσεως. Θα ξεκινήσουμε τον πρώτο γύρο να τα απαντήσουν. Θα ξεκινήσουμε τους συντονιστές. Παρακαλώ τους συντονιστές να παραμείνουν στα χρονικά τους ε, όρια, ο καθένας για δύο λεπτά. Ο Πίτερ Λίζεν είναι πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις εισηγή και ιδιαίτερα για την τελευταία δήλωσή σας για τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και έχω μια ερώτηση, θα ήθελα μια διευκρίνηση. Αναφερθήκατε στην ε, επιστολή την οποία ε, ο πρόεδρος ο ε, Τζοβάνι Λαβία, η κυρία Γκροστέτο και άλλοι συνάδελφοι έστειλαν όπου αναφέρουμε τις ανησυχίες που έχουμε σχετικά με τις εργασίες στο Συμβούλιο και την Κομισιόν σχετικά με την επίτευξη των στόχων ε, για το 2030. Χρειαζόμαστε λοιπόν νέα δομή διακυβέρνηση. Παλιά υπήρχε ένα έγγραφο που έλεγε ότι το Κοινοβούλιο, όπως και άλλοι ενδιαφερόμενοι, άλλοι stakeholders, ε, θα συμμετάσχει. Αλλά αυτό δεν αρκεί για μας. Φυσικά είναι καλό το να συμμετέχει το Κοινοβούλιο, αλλά εάν δεν συμμετέχει ως συνομοθέτης σε μια οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, για παράδειγμα, ε, τότε αρχίζουμε και ανησυχούμε. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο αφορά όχι μόνο τη δική μας Επιτροπή και την Επιτροπή Ήτρε, αλλά το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν ε, μπορώ να φανταστώ εσεί ή ο Ζαν Κλοντ Juncker να μπορέσετε να συμφωνήσετε όλα αυτά τα θέματα να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά σε διακυβερνητικό επίπεδο. Ερώτηση λοιπόν, αναφερθήκατε στο θέμα της ενεργειακής απόδοσης. Ο Ζαν Κλοντ Juncker στην ομιλία του ε, είπε ότι τουλάχιστον 30% δεσμευτικός στόχος ο Άριας Κανιέτε επίσης αναφέρθηκε στο στόχο αυτό. Θα αποτελέσει και αυτό μέρος των προτάσεών σας. Ευχαριστώ πολύ. Ματία Γκέρτα. Ευχαριστώ πολύ, Αντιπρόεδρε. Αναφερθήκατε στους ακρογωνιαίους λίθους για την Ενεργειακή Ένωση. Και μία λέξη που είπατε θα ήθελα να την τονίσω. Είπατε, μιλήσατε για την αξιοπιστία και έχουμε δυσαρεστηθεί με κάποιες ε, δράσεις ή παραλήψεις, ε, την ανάκληση του ενεργειακού πακέτου. Χρειαζόμαστε όμως ε, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία, χρειαζόμαστε συνομιλία όπως εσείς συνομιλείτε μαζί μας. Διότι στο κάτω-κάτω το θέμα είναι πού θα επενδύσουμε. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι δυνατόν να έχουμε ενεργειακή ένωση και θα πρέπει να συλλέξουμε τους απαραίτητους πόρους για κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις παρατηρήσεις σας αυτές και ο συνάδελφος Λίζε μόλις αναφέρθηκε στο ε, μοντέλο διακυβέρνησης, δεν θα αναφερθώ σε αυτό, θα αναφερθώ όμως στον οδικό χάρτη προς το Παρίσι. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα μπορέσετε να παρουσιάσετε το διπλωματικό πακέτο και να διαπραγματευτείτε με πολύ καλό τρόπο. Το θέμα όμως τελικά είναι ποιος έχει την τελική ευθύνη. Καλό θα είναι να την έχει ο ε, αντιπρόεδρος της Κομισιόν, αλλά θα πρέπει οι διεθνείς εταίροι να γνωρίζουν με ποιον διαπραγματεύονται. Κατά τη γνώμη μου, η Ενεργειακή Ένωση συνδέεται στενά με την κλιματική πολιτική, θα πρέπει λοιπόν εδώ να έχουμε ισχυρότερη διασύνδεση ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να γνωρίζουν ε, πώς εργαζόμαστε. Τιμές ε, της ενέργειας. Όταν φτάσουμε σε ενεργειακές τιμές τις οποίες δεν μπορεί να πληρώσει ο ιδιώτης, ε, τότε θα χάσουμε και τα τελευταία ίχνη εμπιστοσύνης των πολιτών. Τίθεται λοιπόν ε, το θέμα της ε, αποπληρωμής ε, των δανείων και των τόκων. Άνθρωποι που δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τον ενεργειακό τους λογαριασμό θα πρέπει να βοηθηθούν με προγράμματα ενεργειακής απόδοσης. Κατά τη γνώμη μου σημαντικό θα είναι για την ανάπτυξη των ανάσχομων πηγών ενέργειας θα είναι να προωθήσουμε διασυνοριακά προγράμματα υποδομών. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται ε, να μην μπορούμε να βρούμε μια ευρωπαϊκή λύση στην ε, χώρα μου ε, έχουμε τέσσερις ε, ζώνες εφαρμογής της ενέργειας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισήγησή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ματίας, η κυρία Κέρλινγκ από το ECR. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Άνετα μπορώ να θέσω το ερώτημά που αφορά το άνοιγμα προς τις ανανεώσιμες. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Κυρίως όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, τη χώρα μου. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες για, χρησιμοποιώντας τα, την παλήρια για την παραγωγή ενέργειας. Και έχουμε φτιάξει στο, στη, στον κόλπο του Σβάνση ε, μια μικρή λίμνη και τελικά θα παράγει ενέργεια που θα ενωθεί με το Εθνικό Δίκτυο του 2018. Αυτό μπορεί να κλιμακωθεί, να κατασκευαστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα και να καλύψει όλα τα Βρετανικά νησιά και ίσως και άλλα μέρη της Ευρώπης να παράγουμε ενέργεια από την Παλήρια. Τεράστιες δυνατότητες υπάρχουν και αυτό το πρόγραμμα ε, προχώρησε με ελάχιστη οικονομική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν αναπτυξιακή τα άλλη. Τι τονίζω. Είναι πόρος όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και για την Ευρώπη. Έχουμε τις μεγαλύτερες παλιροϊκές ροές. Κυρίως εδώ στο Δέλτα που έχουμε φτιάξει αυτό το πρόγραμμα έχουμε τις μεγαλύτερες μεταπτώσεις με την αλλαγή της παλήρειας στον κόσμο. Άρα είναι τεράστια πηγή. Μεγάλες δυνατότητες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Και αυτό το έργο θα κατασκευαστεί κατά 65% στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να παράξουμε τους τροβιλαντιδραστήρες, αλλά τα άλλα μπορούμε. Οι ανανεώσιμες θεωρούνται σαν κάτι παγιωμένο. Ε, πράγματι δημιουργούν πάρα πολλές νέες δυνατότητες. Πώς θα στηρίξετε τις νέες δυνατότητες, τι σχέδια έχετε, πώς θα εξασφαλίσετε ότι η κατασκευή, ε, η ανάπτυξη των ιδεών και η κατασκευή και η υλοποίησή τους θα παραμείνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κ. Φαρία για την Άλτε. Ευχαριστώ. Θέλουμε να έχουμε μια νέα ενεργειακή αγορά Και αυτό είναι παλιά ιστορία, παλιά έμπνευση. Φτάσαμε στο 2015 και εξακολουθούμε να καθορίζουμε, να διαμορφώνουμε στρατηγικές για την επίτευξη του παναφερθέντος στόχου και για τους πολίτες και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική εδώ παρουσία σας κύριε Επιτροπέ. Η ενεργειακή πολιτική σε εθνικό επίπεδο, διάφορες εθνικές ενεργειακές πολιτικές, προστάτευαν εθνικά συμφέροντα. Επικρατούσαν τα εθνικά συμφέροντα και όχι τα κοινά ευρωπαϊκά. Ε, ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση αφορά την αγορά του πετρελαίου. Μιλήσατε για μια μεταρρύθμιση ενεργειακή ενεργειακής πολιτικής στην Ευρώπη, για μια νέα ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη. Ερώτηση. Πώς αξιολογείτε τι διασυνοριακέ διασυνδέσει ε, βάσει των διαφόρων προγραμμάτων για τα κοινοφελή προγράμματα παρακολουθείτε όλος ιδιαίτερο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόοδο που επιτυγχάνεται σε αυτό το τομέα, κυρίως στις απομονωμένες ε, περιοχές και κυρίως στην Ιβηρική Χερσόνησο. Θα υπάρξει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων κάποια παρέμβαση. Η Ευρώπη έχει καταναλώσει ε, πάρα πολύ άνθρακα για την ηλεκτρική ενέργεια, για την παραγωγή της, Βλέπουμε ότι στη ΣΥΠΑ παράγουν φυσικό αέριο από το σχιστόλιθο. Ξέρουμε ότι ο άνθρακος είναι υπεύθυνο για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Περίπου 18.400 άνθρωποι είναι θύματα της ρήπανσης, ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Πολλά δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο δαπανώνται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μπορούν να εσωτερικευτούν αυτά τα αρνητικά στοιχεία κατά κάποιο τρόπο. Κονέτσινα, συνάδελφε. Η κυρία Κονέτσινα. ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, τολμώ να πω ότι κάποιοι συνάδελφοι δεν μπόρεσαν ε, να έρθουν. Δεν, δεν, θέλαμε να σας δούμε, μάλλον θα σας δούμε από κοντά, από παλιά. Σας στείλαμε διάφορες επιστολές και χαίρομαι που είχατε το θάρρος να έρθετε εδώ να συζητήσετε μαζί μας την Επιτροπή μας. Ελπίζω αυτό να συνεχιστεί και την επόμενη τετραετία και να είστε ε, παράδειγμα για τους συναδέλφους σας, τους άλλους επιτρόπους. Έχετε πει επανειλημμένα ότι στα πλαίσια της Ενεργειακής Ένωσης τα προβλήματα είναι η υψηλή τιμή της ενέργειας και ότι πολλά α, νοικοκυριά δεν μπορούν να πληρώσουν τους ενεργειακούς λογαριασμούς τους. Τι θα κάνετε. Είναι εξωθρύνητη αυτή η κατάσταση. Έχετε συγκεκριμένα μέτρα που ετοιμάζετε. Θα ήταν ενδιαφέρον να τα ξέρουμε για τη μελλοντική συζήτηση. Αναφερθήκατε στην Επιτροπή τα αναφέρατε κάποια στοιχεία. Αυτό που μου λείπει είναι ποιοι είναι οι στόχοι, πώς θα υλοποιηθούν οι θεωρίες. Αναφερθήκατε σε οικονομίες. Χρειάζεται σωστή ορθολογική προσέγγιση για την οικονομία. Πώς θα εμποδίσετε τη σπατάλη ενέργειας. Τη σπατάλη της ενέργειας. Πώς θα τη σταματήσετε. Για την ανάπτυξη των διαφόρων δικτύων. Για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. Με τις διασυνδέσεις μεταξύ των δικτύων. Τι θα γίνει σε κάποιες χώρες αναπτύσσονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κολλάει η διαβίωσή του στα σύνορα. Θέλουμε μεγάλα δίκτυα. Ούτως ώστε να μην υπάρχουν οι ελλείψεις ε, ενέργειας και blackout όπως συνέβη στην Τσεχία. Περνάνε τα μεγάλα δίκτυα από την Γερμανία, την Τσεχική Δημοκρατία και αν δεν ανανεωθούν τα μεγάλα δίκτυα μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή, ε, τα καλύτερα, την καλύτερη ενεργειακή ένωση, αλλά ίσως αν δεν υπάρχει σωστή ροή της ενέργειας και ο έλεγχος του ροής της ενέργειας να μένουν κάποια κάτι χωρί ενέργεια. Basic για τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σεύκοβιτς που ήρθατε και που ακούτε τις επιθυμίες του Κοινοβουλίου όσον αφορά την Ενεργειακή Ένωση. Πολύ το εκτιμάμε. Τώρα στη συζήτηση εγώ θα περίμενα. Εδώ είμαι, εδώ είμαι, δεν με έχετε δει. Εδώ είμαι. Ξέρω, είναι μεγάλη αίθουσα και δεν με εντοπίζετε εύκολα. Εδώ είμαι. Λοιπόν, έλεγα να συμφωνήσουμε του πέντε πυλώνε. Μα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Όταν μιλήσει κανεί για του πέντε πυλώνε, ωραία. Φυσική επιλογή. Αλλά τέλη Φεβρουαρίου περιμένω η Επιτροπή να έχει βάλει στην ατζέντα συγκεκριμένα και καυτά θέματα. Γιατί αλλιώς θα μιλάμε για αοριστείες. Γιατί να διαφωνήσουμε. Όχι, πρέπει να βάλετε τα θέματα στο τραπέζι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα μια επιτροπή η οποία λέει ότι θέλει να είναι πιο πολιτική από ό,τι κατά το παρελθόν. Αν αυτές είναι οι προτεραιότητές σας, τότε ελάτε με πολιτικά ζητήματα την επόμενη φορά. Τρία έχω να σας ε, θέσω και θέλω την απόψή σας. Πρώτον, η Ενεργειακή Ένωση πρέπει να ονομαστεί Κλιματική και Ενεργειακή Ένωση. Γιατί αυτό θα είναι το κλειδί στο μέλλον. Πώς θα συνδέσουμε την κλιματική αλλαγή με την ενεργειακή ασφάλεια. Και θα ήθελα αυτή η Επιτροπή να τα συνδέσει αυτά τα δύο που πάνε χέρι-χέρι έτσι κι αλλιώ. Κλιματική και ενεργειακή ένωση. Τότε θα διαπιστώσουμε ότι θα έρθει με πραγματικά δεσμευτικό ενεργειακό πρόγραμμα. Και επιμένω στο δεσμευτικό. Δεύτερον, Λέτε ότι η Επιτροπή Γιούνκερ λέει θέλει να είναι η πρώτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μα πώς γίνεται αυτό όταν έχουμε βγει 5% κάθε χρόνο μέχρι το 2020 και μετά το 2020 θα πέσουμε στο 1% κάθε χρόνο. Αν τηρήσετε το στόχο του 27%. Δεν είναι σοβαρά αυτά αν θέλετε πράγματα να μείνετε πρώτοι. Τρίτον, κάθε χώρα μέλος λέει τα θέματα του, αλλά οι συνθήκε λένε ότι κάθε χώρα μέλος θα έχει το δικό του ενεργειακό μείγμα. Όσο ισχύει αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα λέμε μπλα μπλα μπλα, αλλά πείτε μου, θα αρχίσετε τη συζήτηση εκείνη που θα λέει ότι αυτό το άρθρο πια δεν θα υπάρχει ώστε το κάθε κράτος να έχει το δικό του ενεργειακό μίγμα. Αλλιώς θα επικρατεί αδιαφάνεια και καμία συνοχή. Τέλος, για το EFTD, Τι Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε την Πρόεδρε. Θέλω να επενθυμίσω ότι οι τελευταίοι επιστήμονες έχουν δείξει ότι οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα έρχονται από τα ορυκτά και είναι κάτι ασύμβατο με τον στόχο μας να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους δύο βαθμούς. Τα ξέρουμε αυτά σε διεθνές επίπεδο. Το 1 τρίτο είναι πετρέλαιο, τα αποθέματα του φυσικού αερίου και του άνθρακα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, πρέπει να παραμείνουν στο υπέδαφος μέχρι το 2050 αν θέλουμε πράγματι να περιορίσουμε την άνοδο της θερμοκρασίας κάτω από τους δύο βαθμούς στον πλανήτη μας. Διάβασα την πρόταση που λέει ότι πρέπει να μοιραστούμε τους πόρους μας, να συμπληρώσουμε τις υποδομές μας και να ενώσουμε τις δυνατότητές μας με τις τρίτες χώρες, λέτε. Είμαι μέλος και στην Επιτροπή για τις σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ. Υπάρχει ψήφισμα που έχουμε ψηφίσει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου επιμένουμε για τις ε, πηγές αυτές του υπεδάφους και στην Ευρώπη και στην Αφρική και θέλουμε να μειώσουμε την εκμετάλλευση των πόρων αυτών στην Ευρώπη αλλά να τις αυξήσουμε στην Αφρική δηλαδή άνθρακας, πετρέλαιο κλπ. Δεν θα ρηπαίνουν πια την Ευρώπη, θα ρηπαίνουν όμως την Αφρική. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια στάση υποκριτική. Το λόγο έχει τώρα ο Αντιπρόεδρος Σεφκοβιτς για το να απαντήσει στον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση του κύριου Λίζερ, που ήταν για τη διακυβέρνηση. Θα μιλήσω λίγο παραπάνω για αυτό το ζήτημα, γιατί ξέρω ότι ενδιαφέρει τους περισσότερους από εσά. Το πρώτο που πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι χρειαζόμαστε μια εύρωστη διακυβέρνηση για να γίνει η πραγματικότητα η Ενεργειακή Ένωση και να πετύχουμε τους στόχους μας για το 2030. Τι πρέπει να καλύπτει αυτή η διακυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα θα μας επιτρέπει να έχουμε πιο συνεκτικές πολιτικές. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για να αυξήσουμε και την προβλεψιμότητα. Μια προϋπόθεση για να έχουμε μεγάλες επενδύσεις στην Ευρώπη. Όταν μιλάμε με επιχειρηματίες και επενδυτές και εσείς τα ξέρετε, το πιο βασικό για να επενδύσουν στις ανώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. είναι να υπάρχει ένα ρυθμιστικό σταθερό πλαίσιο. Αυτό είναι που θα κάνει το θαύμα, που θα διασφαλίσει ότι οι πολιτικές μας θα παραμείνουν εφόσον υπάρχουν επενδύσεις και θέλουμε να γίνουν επενδύσεις στις προοδευτικές τεχνολογίες του μέλλοντος. Αλλά γι' αυτό πρέπει να έχουμε ρυθμιστική σταθερότητα. Αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο σύστημα διακυβέρνησής μας. Δεύτερον, πρέπει να αναπτύξουμε ένα σύστημα διακυβέρνησης που θα μας επιτρέψει να δώσουμε κίνητρα στην περιφερειακή συνεργασία. Να αποφύγουμε κάποια παραδείγματα που είχαμε και φάνηκε στον πρώτο γύρο ερωτήσεων όταν εκπλήσουμε τους γειτονές μας, δεν τους μιλάμε και απλώς τους βάζουμε μπροστά στο τετελεσμένο. Είναι κάτι που οδηγεί τα ενεργειακά τους δίκτυα την οικονομία τους σε δύσκολη κατάσταση. Και βέβαια κάτι πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η διακυβέρνηση αυτή να μας επιτρέψει να πετύχουμε τους στόχους που έθεσε τον Οκτώβριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή τουλάχιστον 40% που είναι δεσμευτικός όρος για το διοξίδιο του άνθρακα. Και τουλάχιστον θα έλεγα 27% ανανεώσιμες. Πάλι πρόκειται για δεσμευτικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τουλάχιστον 27% ενεργειακής απόδοσης που ήταν ένα συμβατικό μέτρο, ενδεικτικό στόχος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως και τον τέταρτο στόχο που έχει να κάνει με την σύνδεση 50% διασύνδεσης στην Ευρώπη μέχρι το 2030. Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς όμως εννοείται ότι χρειαζόμαστε νομοθεσία. Άρα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα ETS, εμπορία ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Να έρθουμε με προτάσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσει και στον τομέα που δεν εμπίπτει στο σύστημα ETS να δούμε την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, για τα κτίρια, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ. κλπ. Συνεπώς, όλα αυτά είναι φιλόδοξη νομοθετική στόχη που έχουμε στην ατζέντα μας. Και σαν πακέτο πρέπει να δούμε την Ενεργειακή Ένωση, γιατί στα τέλη του Φεβρουαρίου αυτό που θέλουμε να σας φέρουμε είναι το κείμενο για την Ενεργειακή Ένωση που να περιγράφει λεπτομερώς πώς θα πετύχουμε τη μετάβαση αυτή, την αλλαγή αυτή. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει και ένας χάρτης πορείας που θα τα συνοδεύει όλα αυτά με συγκεκριμένες δράσεις για να οικοδομηθεί η Ενεργειακή Ένωση. Θέλουμε επίσης και κάτι ξεκάθαρο για το πώς θα ελέγξουμε καλύτερα τις υποδομές. Κάποιοι ευρωβουλευτές με ρώτησαν γι' αυτό πώς θα έχουμε καλύτερες διαδικασίες ελέγχου, ε, προτεραιοτήτων, όσον αφορά τις υποδομές, προγράμματα για υποδομές που πραγματικά να συνεισφέρουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο σε περιφερειακό ή σε εθνικό. Θέλουμε να συνδέσουμε επίσης το πακέτο για την Ενεργειακή Ένωση με τον χάρτη πορείας εν του Παρισιού. Τι διπλωματική επιρροή θα προσπαθήσουμε να έχουμε μέσα στους επόμενους μήνες εν του Δεκεμβρίου του Παρισιού. Και το όλο πακέτο πρέπει να συμπληρωθεί με τις ανακοινώσεις για το 10% για τις διασυνδέσεις. Βλέπετε πολλά σας, θα σας φέρουμε το Φεβρουάριο. Και όλο αυτό το νομοθετικό έργο εννοείται συμπεριλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο ρόλος σας είναι ζωτική σημασία. Θα συμμετέχετε στην όλη διαδικασία και θα συνεργαζόμαστε στενά. Ένα ακόμα ζήτημα που προσπαθούμε να αλλάξουμε είναι το εξή. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία για το τι γίνεται εν ώψη των στόχων του 2030 κλπ. Η Ενεργειακή Ένωση πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι, είπατε, με την κλιματική αλλαγή. Ναι, άρα χρειαζόμαστε ένα σύστημα, έναν κύκλο όπου θα μπορούμε να βλέπουμε όλες αυτές τις πτυχές από μία οπτική γωνία και να μπορούμε έτσι να έχουμε μια συνολική εικόνα και συζητήσεις και διμερώς αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σας και με το Συμβούλιο να ξέρουμε συνολικά πώς προχωράμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε ένα σύστημα λοιπόν παρακολούθησης και αναφοράς με την αναγκαία ευελιξία που να μας επιτρέπει να καταλήγουμε σε συγκεκριμένες ιδέες για το πού μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, πού μπορούμε να δώσουμε κίνητρα στις χώρες μέλη να κάνουν περισσότερα και σε τι βαθμό μπορούμε να τους επικρίνουμε ότι δεν κάνουν αρκετά. Αυτές είναι οι βασικές ιδέες. Θα είναι πιο συγκεκριμένες το Φεβρουάριο όταν θα έχουμε εγκρίνει το πακέτο για την Ενεργειακή Ένωση και πώς θα το εφαρμόσουμε. Εννοείται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει πλήρως στην όλη αυτή διαδικασία. Επιτρέψτε μου τώρα να κάνω και ένα σχόλιο μετά από αυτά που είπε η κυρία Γκροστέτ για το πακέτο για τα απόβλητα. Στο πακέτο μας για την Ενεργειακή Ένωση θα βρείτε και ένα κατάλογο προτεραιοτήτων, δράσεων κατά προτεραιότητα. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια νέα πρόταση, πιο φιλόδοξη που θα εξετάζει ολόκληρο τον κύκλο των προϊόντων. Όχι μόνο από τη στιγμή που αρχίζει να χρησιμοποιείται μέχρι τη στιγμή που το πετάμε το προϊόν, αλλά τον πλήρη κύκλο του που αρχίζει από τη χρήση των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων για να κατασκευαστεί, να συσκευαστεί, να μεταφερθεί, να πεταχτεί και να ανακυκλωθεί. Πρέπει να δούμε πώς αυτή την ανακύκλωση των πρώτων υλών μπορούμε να την διοχετεύσουμε στην ευρωπαϊκή οικονομία να μειωθούν οι μεταφορές. και να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Με εξέπληξε όταν κοίταξα τα ποσά όταν μεταποιούμε το αλουμίνιο πόσο πολύ κερδίζουμε σε ενέργεια. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται από την εξόριξη μέχρι το τέλος στον κύκλο ζωής του αλουμινίου που μπορούμε να εξοικονομήσουμε. Να δούμε λοιπόν την κυκλική οικονομία και την διαχείριση αποβλήτων στο μέλλον. Ο κύριος Βρότο επίσης αναφέρθηκε και στο θέμα του ηλεκτρισμού στη Γερμανία, αλλά όχι μόνο. Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Είμαστε σε ένα τέτοιο επίπεδο κατακαιρματισμού της αγοράς ηλεκτρισμού που χρειαζόμαστε μια νέα αγορά ηλεκτρισμού. Αυτή πρέπει να σχεδιάσουμε και αυτό θα σας προτείνουμε. Να αλλάξουμε την αγορά ηλεκτρισμού. Να ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα, να ανταποκρίνεται στη σημασία που έχουν ενώσιμε πηγέ ενέργεια, να ανταποκρίνεται στι ανάγκε, καλύτερη συνεργασία σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί μόνο μέσα από ένα νέο σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρισμού μπορούμε να πετύχουμε τους σημαντικούς στόχους που έχουμε θέσει στους αυτούς μας. Η κυρία Γκέρλινγκ ρώτησε για τη στήριξη των νέων και προοδευτικών τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας. Η περισσότερη στήριξη στην έρευνα και την ανάπτυξη. Ναι, όπως το προτείνετε πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο και είναι προς το συμφέρον των επιστημόνων. Είναι επίση προς το συμφέρον εκείνων που θέλουν να συγχρηματοδοτήσουν τέτοια προγράμματα στο μέλλον και να μπορούν έτσι να έχουν βοήθεια από το επενδυτικό πακέτο Juncker. Οι αρχικές εκτιμήσεις για τις επενδύσεις αυτές είναι ότι θα κατανεμηθούν 20-27% θα πηγαίνουν στις υποδομές, 27% στις μεταφορές. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την χρηματοδότηση πολλά υποσχομένων προγραμμάτων που είναι σημαντικά για το μέλλον και που μπορεί και οικονομικά να είναι πολύ εύρωστα, επιχειρηματικά. Ο κ. Βάριο ρώτησε πώς θα διαχειριστούμε καλύτερα τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τα TEN. Έχουμε από τα διευρωτικά ταμεία, άλλη χρηματοδότηση είναι από το Connecting Europe Facility, τη διευκόλυνση αυτή συνδέοντας στην Ευρώπη δηλαδή. Έχουμε χρηματοδότηση επίσης, υπάρχει το PCI, που συνδέεται με την στρατηγική του ενεργειακού τομέα και έχουμε και νέες προτάσεις για προγράμματα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το επενδυτικό πακέτο Juncker. Πρέπει λοιπόν να γίνει καλύτερη διαχείριση όλων αυτών των προγραμμάτων, να τα βάλουμε κατά προτεραιότητα, να τη ιεραρχήσουμε δηλαδή και να προωθήσουμε τα προγράμματα εκείνα τα οποία προσφέρουν περισσότερη προστεθέμενη αξία στην Ευρώπη. Αλλά πρέπει να υπάρχει και μία παρακολούθηση στη συνέχεια στις χώρες μέλη. Να δούμε, προχωράνε, αν δεν προχωράνε τότε γιατί να ξοδέψουμε χρήμα, χρόνο και ενέργεια για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν προχωράει. Πρέπει να υπάρχει και παρακολούθηση δηλαδή στη συνέχεια και ενδεχομένω να δικατασταθεί ένα πρόγραμμα που δεν προχωράει από κάποιο άλλο ή να μειωθούν τα χρήματα διδατικών ταμείων ή να χαθούν. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τρόπους με τους οποίους θα παρακολουθούμε την δημιουργία δικτύων και τα προγράμματα που θα χρηματοδοτούνται. Η κυρία Κόνιτσνα αναφέρθηκε στις υψηλές τιμές ενέργειας. Μέρος της αγοράς ηλεκτρισμού είπαμε ότι πρέπει να ανασχεδιαστεί. Και ένα από τα στοιχεία αναθεώρησης θα είναι η ηλιανική τιμή. Γιατί αν δείτε πόσο κοστίζει ο ηλεκτρισμός, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εντάξει είναι διαφορετικά βέβαια από τη, στην Αμερική, αλλά εμείς βάζουμε κόστος μεταφοράς, φόρους και ένα σωρό που αυξάνουν επί δύο, επί τρία την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας εδώ από ό,τι είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Άρα και εδώ πρέπει να έχουμε ειλικρινή συζήτηση και να δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε καλύτερα τις τιμές και να χρησιμοποιήσουμε και καλύτερα τις κατευθυντήριες γραμμές για να περάσουν οι ανανόσιμες πηγές ενέργειας στην πράξη και οι τιμές μας να είναι πιο λογικές και καλύτερες για τις επιχειρήσεις μας. Όσον αφορά τώρα την ε, ενέργειας πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για τον οικολογικό σχεδιασμό και την οικολογική σήμανση προϊόντων. Πολύ συχνά ο τύπος επικρίνει. Εμείς όμως ξέρουμε ότι ο οικοσχεδιασμός είναι πολύ σημαντικός. Αν δούμε τις προσπάθειες που κάνουμε για την ενεργειακή απόδοση, τα μισά αποτελέσματά μας είναι χάρη σε αυτή την νομοθεσία. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι στόχοι για το 2020 επιτυχάνονται χάρη ακριβώ σε αυτήν την οδηγία. Θα εξοικονομήσουμε το ίδιο ποσό ενέργειας που θα μπορούσαμε σε ένα χρόνο. Και μπορούμε φυσικά να αναβαθμίσουμε, να εξυγχρονίσουμε το eco τον οικοσχεδιασμό. Οι πολίτες, οι καταναλωτές θέλουν να ξέρουν ποια είναι η ενεργειακή απόδοση. Είναι λοιπόν πολύ καλό και για την εξοικονόμηση ενέργειας και για μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Να δούμε τώρα την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Εδώ θέλουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αναπτύξουμε κάποιο μέσο το οποίο να επιτρέπει στους Δήμους να είναι πιο θαραλέοι, πιο τολμηροί και να αρχίσουν νέα προγράμματα για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Φυσικά, απλοποιώντας, θα μπορούσε να ήταν απλό. Να, ο λογαριασμός και να χωρίσουμε το κόστος στην επένδυση και στο κτίριο. Μπορούν δηλαδή να υπάρξουν πιο καινοτόμες λύσεις. Στον κύριο Ικχάουτ τώρα. Μερικώς απάντησα ότι δεν πρόκειται μόνο για λόγια, θα υπάρχει συγκεκριμένο πρακτικό σχέδιο για το πώς θα οικοδομήσουμε την ενεργειακή αυτή ένωση. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις ή για νέα νομοθεσία ή για αναθεώρηση της παλιάς νομοθεσίας, προσθέτοντας πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία θα έχουμε και εμείς στη προπτευτική μας θέση εν ώψη του Παρισιού. Όπως αντιλαμβάνεστε, επ' αυτού πρέπει να δουλέψουμε πάνω στα πεσεφωνημένα. Υπάρχει συμφωνία με τις χώρες μέλη μετά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Αυτή θα είναι λοιπόν η βάση για την προπαρασκευαστική μας δουλειά εν ώψη των προτάσεων που θα παρουσιάσουμε με το πακέτο του Φεβρουαρίου. Η τελευταία ερώτηση ήταν από τον κύριο Πεντιτζίνη όσον αφορά τις τιμές του άνθρακα και πώς θα καθοριστούν. Η τιμή του άνθρακα αυτή τη στιγμή δεν είναι κατάλληλη. Το σύστημα ETS δεν λειτουργεί καλά. Πρέπει να έχουμε σταθερότητα στην αγορά πρώτα απ' όλα. Έχω κάποιες ιδέες πώς μπορούμε να συμφιλιώσουμε τις θέσεις των Ευρωβουλευτών της δικιάς σας Επιτροπής και της Επιτροπής Ήτρε με τριμερή διάλογο ελπίζω ότι θα επιτευχθεί συμφωνία. Η Προεδρία είναι προετοιμασμένη. Πολύ σύντομα θα υπάρχουν οι προτάσεις μας για το ETS. Αυτό είναι αναμενόμενο από τη δικιά μας την πλευρά για να βοηθήσουμε στις διαπραγματεύσεις και στο Παρίσι και αλλού. αν υπάρξουν καλά σημάδια θα δείτε ότι και το σύστημα θα λειτουργήσει και πολλά από τα προβλήματα που συζητάμε τώρα θα έχουν εξαφανιστεί εφόσον το σύστημα λειτουργήσει και πάλι ικανοποιητικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς για αυτή την πρώτη ομάδα απαντήσεων. Μπαίνουμε στο δεύτερο γύρο. Παρακαλώ συνάδελφοι να τηρήσετε το χρονοδιάγραμμα. 1,5 λεπτό. Η κυρία Γκροστέτ. Είναι η πρώτη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αναφερθήκατε προηγουμένως στην ενιαία ενεργειακή αγορά. Είπατε ότι θέλετε να αναπτύξετε τη διαδικασία των εφιών πόλεων. Είναι σημαντικό λοιπόν οι Δήμοι να μπορούν να αναπτύξουν νέες αποδοτικές υπηρεσίες, μεταφορές για την ευφυή κινητικότητα, την αξιοποίηση των αποβλήτων, ενεργειακή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Όσον αφορά το δημόσιο φωτισμό, τα κτίρια θα πρέπει να γίνουν ευφυή. E. Θέλουμε ε, καλύτερη διαχείριση της ενέργειας. Πρέπει όμως αυτή η πολύ ωραία ιδέα να μην παραμείνει κάτι τέτοιο. Γνωρίζετε πολύ καλά, για να υλοποιηθούν αυτά χρειάζονται χρήματα. Τι θα κάνετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο γι' αυτό, κύριε Επίτροπε, Πώς θα συνοδεύσετε αυτή την ανάπτυξη των νέων ευφυών δικτύων. Γνωρίζετε επίσης ότι η τοπική αυτοδίκηση αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες σήμερα για να καλύψει τα κενά του προπολογισμού. Άρα πρέπει να στηρίξετε δημόσια, την τοπική αυτοδίκηση. Τι θα κάνετε λοιπόν για αυτές τις ευφυείς πόλεις. Ευχαριστώ. Ο κ. Παουλούτσι έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, η δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης αν θέλουμε να αποφύγουμε θεωρίες, θεωρητική συζήτηση, περνάει και από την υπέρβαση των στρεβλώσεων της εσωτερικής αγοράς μεταξύ χωρών. Όσον αφορά τους κανόνες, οικονομικές ενισχύσεις και πολιτική στήριξη γενικά. Να προσέξετε και το εξή. Το ETS είναι ένα από τα ισχυρά σημεία των διαφορών πολιτικών που ακολουθούμε για την καταπολέμηση αλλαγή του κλίματος ε, και για τη δημιουργία της εταιρικής αγοράς. Πώς θα άρθρο Έξι, Προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα για το ETS, για τι επιχειρήσει στον τομέα για να αποφευχθεί η διαρροή του άνθρακα, για να αντισταθμιστούν οι δαπάνε των εκπομπών. Τι έγινε στη Χαλιβουργία, Φερρυπίν. Κάποιε χώρε ε, επέβαλαν τα μέτρα στι επιχειρήσει, άλλε όχι. Οπότε υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Διαφορετική εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων του ETS στι χώρε τη Ευρώπη. Αυτή η διαφοροποιημένη εφαρμογή επέφερε ενδοκινοτική στρέβλωση. Και ανάλογα με τους εθνικούς υπολογισμούς γίνεται διανομή των δικαιωμάτων. Υπάρχει ανισότητα και επηρεάζεται και το ΑΕΠ των χωρών. Ε, άμα κάποιες χώρες συμμορφώνται και κάποιες όχι. Δεν πάει η κατάσταση. Μέσω ψηφίσματος του Δεκεμβρίου το Κοινοβούλιο έχει τοποθετηθεί ήδη. Η αναθεώρηση του ETS δεν αναφέρεται στις ιδιαίτερες, στις ειδικές αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να καλυφθούν αυτές οι στρεβλώσεις. Πώς θα προχωρήσετε μέσω κάποιας αναδιαμόρφωσης των ε, διατάξεων του ETS για να μην υπάρχουν αυτές οι στρεβλώσεις. Ευχαριστώ, η κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ. Θέτω το ερώτημα εκ μέρους του κυρίου Ντόνκεν που εκφράζεται εκ μέρους της ομάδας μου στην Επιτροπή για την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος. Και λέει, όπω γνωρίζετε, το δίκτυο τη Βόρεια Θάλασσα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην Ενεργειακή Ένωση. Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει ενεργειακέ ροέ σε διάφορε χώρε και μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη όπω το Ηνωμένο Βασίλειο να εξαγάγουν περισσότερη ενέργεια από αυτή παράγουν. Μπορείτε να μα διαβεβαιώσετε ότι το δίκτυο τη Βόρεια Θάλασσα θα έχει προτεραιότητα στο σχεδιασμό σα για την Ενεργειακή Ένωση και θα δεσμευτείτε να δημοσιεύσετε πλήρη έκθεση όσον αφορά την πρόοδο πριν το τέλο Σεπτεμβρίου ούτως ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε την όλη κατάσταση του προγράμματος και να εστιαστούμε επί της υλοποίησης του προγράμματος ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Μέιστερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, και εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση του προγράμματός σας. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις έχω. Η μία σχετίζεται με την Ενεργειακή Ένωση και την Ενεργειακή Υποδομή. Ο κύριος Τένιερ είπε ήδη πριν από εσά ότι είναι σημαντικό να οικοδομήσουμε την υποδομή στην Ευρώπη ώστε να μπορέσουμε να συνδέσουμε τον άνεμο του Βορρά και τον ήλιο του Νότου. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, έχετε συνομιλίες με τα κράτη-μέλη για την καλύτερη εφαρμογή αυτής της ιδέας. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη συνδέεται με την ξυλία ως πρώτη ύλη. Ιδιαίτερα στον βορρά της Ευρώπης υπάρχει ε, πολλή ξυλία, αλλά και όσον αφορά το οικολογικό αποτύπωμα, η ξυλία έχει πολύ καλύτερη βαθμολογία από τον Χάλιβα, για παράδειγμα. Θα ήταν δυνατόν λοιπόν να τονίσουμε περισσότερο την χρήση της ξυλίας στις κατοικίες, όχι μόνο για τους αλλεργικούς, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω εάν το έχετε λάβει υπόψη αυτό στην γενική εξίσωση που αφορά την ενέργεια και την ενεργειακή κατανάλωση και παραγωγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σιωριστή. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και τον αντιπρόεδρο Ομολογώ ότι καλή μουσική ακούγεται στα αυτιά μου όλα αυτά που μας είπατε. Αλλά όταν φτάνουμε στην πραγματικότητα, στο ρεαλισμό και όχι μόνο στα σχέδια, Μιλάτε για περισσότερες ανανεώσιμες, μιλάτε για ενεργειακή απόδοση, που, ότι τα παιδιά μας δεν θα πληρώνουν τα λάθη που έχουμε κάνει εμείς προηγούμενοι. Εννοείται ότι συμφωνώ, αλλά διαβάζω και νέα για το για το σχιστολιθικό αέριο και την ε, ρογμάτωση. Εκατομμύρια γη χάνεται. Κατά τη γνώμη μας όλα αυτά θα διευκολύνουν απλώς και μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις που θα εκμεταλλεύονται τους μικρούς. Εγώ ανατριχιάζω όταν σας ακούω λοιπόν για αυτά. Και έπειτα είπατε ότι βασίζεστε στους δήμους, στους πολίτες. Στη χώρα μου τουλάχιστον, ακόμα και στο χωριό από που εγώ, που είναι ένα μικρό, δεν υπάρχει τέτοια επαφή. Ούτε ενημερωνόμαστε, ούτε γίνονται μελέτες για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στη δημόσια υγεία από τις μεγάλες επιχειρήσεις fracking, ρογμάτωσης. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά οι συνέπειες είναι πράγματα που πρέπει να ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλω την απόψή σας επ' αυτού. Thank you very much. And now Mr. Turmes. Ε, thank you. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Union ε, can be... Η Ενεργειακή Ένωση μπορεί να είναι επιτυχής. Αυτό πιστεύω. Πρέπει όμως να έχουμε κάποια ορατά προγράμματα το δίκτυο της Βόρειας Θάλασσας αναφέρθηκε. Εγώ ζητώ έναν πόρο για 50 δισεκατομμύρια για αυτό το σκοπό. Αναφέρατε ευφυείς πόλεις. Πόλεις που θα είναι πιο κοντά στους πολίτες. Μια πτυχή είναι αυτή. Η ενεργειακή πολιτική μας να είναι πιο ορατή. Μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων. Δεύτερο ζήτημα. σύγκληση των ενεργειακών πολιτικών για την αποδοτική χρήση της ενέργειας στα διάφορα κράτη-μέλη. Τρεις οδηγίες υπάρχουν και προσπαθούν να πετύχουν τη σύγκληση. Η οδηγία την ανανεώσιμη ενέργεια φέρνει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Και έχουμε διάφορες ομάδες που επικρίνουν το κόστος των εθνικών μέτρων στήριξης. Αυτό δεν στηρίζεται επιστημονικά ανακατεύουν στη μελέτη που παρουσίασαν στον Ταβός ε, διαφορετικά πράγματα, ανάμεικτα. Οι ανανεώσιμες μπορούν να κάνουν πολλά και θα έπρεπε να συνεχίσουμε τη θέσπιση συνεχιζό, ε, σχετικής νομοθεσίας. Θέλουμε νομοθεσία για την κατασκευή αποδοτικών κτηρίων και νέα γενιά ε, οδηγιών για τα κτίρια διότι πρέπει να ανακαινιστούν, να ανανεωθούν τα κτίρια της Ευρώπης. 80% συν των ε, κτιρίων ε, πρέπει να ανανεωθούν. Και η οριζόντια οδηγία για την αποδοτική ε, χρήση της ενέργειας προβλέπει κάποια πράγματα στην, στο άθρο 7. Χρειαζόμαστε οικολογική κατασκευή κτίριων. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι για σας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αυτή νομοθεσία που είναι και ο μόνος τρόπος να παίξει ρόλο το Κοινοβούλιο. Θα ακολουθήσει σωστή πορεία. Αλλιώς θα παραμεριστούμε. Μήπως τελικά δεν ακολουθείτε τους Βρετανούς που δεν θέλουν νομοθεσία πάνω σε αυτά τα θέματα μετά το 2020. Ευχαριστώ και ο Ματζουρόνης έχει το λόγο. Ευχαριστώ. όσον αφορά την Ενεργειακή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση, αυτή η Ένωση μας εγγυάται την ενεργειακή ανεξαρτησία. Κάτι πολύ σημαντικό, εν ώψη απρόβλεπτων μονοπωλίων εφοδιασμού ενεργειακού και μεγάλης εξάρτησης από χώρες όπως είναι η Ρωσία. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να εξασφαλίσουμε ενεργειακή και οικολογική ασφάλεια. Έχω την εξή ερώτηση. Πώς θα ενθαρρύνετε την πράσινη ανάπτυξη, πώς θα εξασφαλίσετε μακροχρόνια ανάπτυξη ανανεωσίμων πηγών ενεργείας, ποιες υποχρεώσεις θα προβλέπονται ούτως ώστε να μειωθεί η εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να ενθαρρυνθεί η τοπική χρήση ενεργειακών πηγών, μάλλον η χρήση τοπικών ενεργειακών πηγών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάλτσο έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. δεν μας μιλήσατε για τη Μόσχα. Συναντήσατε εκεί τον Υπουργό Ενέργειας και τον Πρόεδρο της Γκάσπρομ ε, Και ξέρουμε ότι μέσω πρόθεσμα δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το φυσικό αέριο από την Ρωσία όσον αφορά την ε, ενεργειακή ασφάλεια. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαφοροποιήσουν την, ε, τον ενεργειακό εφοδιασμό τους. Το θέμα είναι τι γίνεται και με τον νότιο διάδρομο, το South Stream. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι εσείς πώς βλέπετε τον αγωγό North Stream όπου θα έχουμε ρωσικό αέριο κατευθείαν προς ε, την Ρωσία με συμμετοχή των Ρώσων κατά 49%. Και επίσης, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει αγωγό στην Τουρκία. Βρίσκεται ρεαλιστικό το πρόγραμμα αυτό. Ε, από τον αγωγό αυτό θα πρέπει να εφοδιάσει η Ευρώπη. Πώς το βλέπετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριο κύριος Ιβομπέλετ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, εδώ είμαι δεξιά. Μπροστά, μπροστά, δεξιά. Ερώτηση Ολλανδιστή. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Πρόκειται για έναν από τους πυλώνες, όπως τον αναφέρετε, της ε, ε, απάλληψης του άνθρακα από το πακέτο Πρόκειται επίσης για την τιμή του ανθρακά και για μια σωστή ισορροπία. Από τη μια μεριά να υπάρχει ένα φιλόδοξο σύστημα ETS με την μεταρρύθμισή του κτλ. Και από την άλλη μεριά πώς να έχουμε χαμηλές τιμές ενέργειας για τις επιχειρήσεις. Πρέπει να δούμε το κόστος της ε, μεταρρύθμισης αυτής. Ποια ε, θα είναι, το έμεσο κόστος ενός μεταρρυθμισμένου συστήματος ETS εθνικό επίπεδο πώς θα υπάρχει η αντιστάθμιση με τι προτάσεις. Πολλοί εδώ πέρα λένε ότι χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό αναρμονισμένο σύστημα για να αποφύγουμε να υπάρχουν ανισότητες σε εθνικό επίπεδο. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό. Και τώρα ο Αντιπρόεδρος ο κύριος Πότ. Πράγματι, για πραγματική ενεργειακή ένωση υπάρχει μια προϋπόθεση. Διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα. Είναι η βάση για τα πάντα. Μπορούμε να συζητούμε ό,τι θέλουμε, αλλά αν δεν έχουμε αυτό το δίκτυο δεν έχουμε τίποτα. Για να υπάρξει το δίκτυο χρειαζόμαστε πραγματικά μια κοινοτική προσέγγιση, συνεργασία κρατών μελών. Μέχρι τώρα σταματά αυτή η πολιτική στα εθνικά σύνορα. Στα σύνορα μεταξύ χωρών, όπως τα, μεταξύ βαλτικών χωρών, μεταξύ Ισπανίας, Γαλλίας κλπ. είναι δύσκολη διασύνδεση η ενεργειακή. Χρειαζόμαστε κάτι ίσως εντελώς καινούριο για να πείσουμε τα κάτι μελη για την ανάγκη, της κοινοτικ... ανάγκη κοινοτικής προσέγγισης. Η ερώτηση είναι πολιτικής φύσεως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάτι καινούριο, εντελώς καινούριο, να πείσει τα κράτη-μέλη, να στηρίξουν την ιδέα. Η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασκήσει μεγαλύτερες πιέσεις. Δεν, έχουν, δεν είμαστε σίγουροι, διότι έχουν αποσυρθεί διάφορα πακέτα από το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω πολιτικών πιέσεων από πλευράς κρατών μελών. Γι' αυτό κάνω και αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Βυζνιεύσκα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να επανέλθω στην ερώτηση που έθεσα κατά την ακρόασή σας. Δεν μου απαντήσατε όμως. Αναφέρομαι στον ρόλο του άνθρακα το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο μακροπρόθεσμα δηλαδή, καταρχάς μέχρι το 2300, αλλά και πιο μακροπρόθεσμα στο το 2050. Θεωρείτε ότι οι χώρες που χρησιμοποιούν άνθρακο όπως είναι η Πολωνία θα πρέπει να έχουν επαρκή ευελιξία ώστε να έχουν ενεργειακό μείγμα χωρίς κοινωνικούς κινδύνους και κοινωνικό κόστος ή θα εισαχθεί η μεταρρύθμιση χωρίς μεταβατικό στάδιο και η Πολωνία ε, έχει πολύ άνθρακα. Θα είναι πολύ δύσκολη για αυτήν η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Πόσο μάλλον υπό το φως όσων συμβαίνουν στην Ουκρανία. Θα ήθελα να αναφερθείτε και στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές ε, που αναφέρατε ως έναν από τους πυλώνας της Ενεργειακής Ένωσης. Πώς θα διατηρήσουμε θέσεις απασχόλησης στον ε, τομέα των ανθρακοριχείων και η Ευρωπαϊκή Ένωση πώ θα μπορεί να βρίσκεται επικεφαλής στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Μέλλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την παρουσία του εδώ. Στο τελευταίο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έγινε λόγος περί Τυχών που συνδέονται με την Ιβυρική Χερσόνησο και σχετικά με την ενέργεια. Καθορίστηκαν στόχοι σχετικοί στο Συμβούλιο. Ερώτηση, τι προτίθεστε να κάνετε συγκεκριμένο, ούτω ώστε να ληφθούν υπόψη αυτά που υπόθηκαν. Και θα ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση, διότι η Ιβυρική Χερσόνησος έχει 7 από τα 12 τερματικά του υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή οι διασυνδέσεις μεταξύ Βυρικής Χερσονήσου με τη Γαλλία δεν ξεπερνούν το 1,6%. Να υπενθυμίσω κύριε Επίτροπε ότι κάποια κράτη-μέλη εξαρτώνται τώρα 100% από τη Ρωσία για την κατανάλωση φυσικού αερίου και για τον ενεργειακό τους εφοδιασμό. Συνεπώς θα πρέπει πραγματικά να προβληματιστούμε από αυτού. Δεν είναι έξυπνη αυτή η μεγάλη εξάρτηση από τη Ρωσία. Λοιπόν, μία παρέμβαση στην Ιβηρική Χερσόνησο θα μειώσει αυτή την εξάρτηση. Τι θα κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σεβαστεί αυτή την πτυχή, ο κύριος Λάινεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, η Ενεργειακή Ένωση φαίνεται θα είναι μια αποστολή πάρα πολύ δύσκολη, σχεδόν αδύνατη με 28 διαφορετικά κράτη-μέλη. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου τις μεταρρυθμίσεις στην ενεργειακή αγορά και πώς μπορούμε να αποφύγουμε φαινόμενα lock-in, δηλαδή μια εκμετάλλευση που ξεκινάει τώρα να επιμείνει να λειτουργεί επί 50 χρόνια. Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό έχοντας ε, το βλέμμα μας στο 2020 το 2030. Και όσον αφορά τους αγωγούς, τι είναι απαραίτητο, τι είναι περιττό. Και τελευταία παρατήρηση, αναφερθήκατε στην τοπική παραγωγή ενέργειας και η κυρία Γκροστέτα αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας καλέσω να συνεργαστείτε εντατικά με αυτό το επίπεδο, διότι υπάρχουν ε, εδώ πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης της ενεργειακής πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σουίτσα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την παρουσία του εδώ σήμερα. Ξέρουμε ότι η ενέργεια από την Ανατολή στοιχίζει πολλά και οικονομικά και πολιτικά και ως Ένωση θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις πηγές μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα αυτόν. Στις διαφάνειες που μας δείξατε, αναφέρατε τα 28 διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένης της Κροατίας, της πατρίδας μου, με βάση όμως τις συνθήκες τα κράτη-μέλη μπορούν να επικαλεστούν ρήτρα που να λέει ότι αποφασίζουν τα ίδια για το ενεργειακό τους μείγμα. Υπάρχουν χώρες όπου υπάρχουν ποσοστώσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αποτελούν την... το βασικό πρόσκομα για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας αναφερθήκατε στα δίκαια, αναφερθήκατε και στην ε, νομοθετική σταθερότητα, την ρυθμιστική σταθερότητα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς ε, σκοπεύετε να εφαρμόσετε αυτήν τη σταθερότητα, διότι χωρίς αυτήν θα είναι αδύνατον να εφαρμόσουμε την Ενεργειακή Ένωση. Πώς μπορούμε λοιπόν να πετύχουμε τέτοια σταθερότητα και φυσικά σε συνεργασία με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό παρά το άρθρο της συνθήκης που λέει ότι τα κράτη-μέλη αποφασίζουν μόνο τους για το ενεργειακό τους μείγμα. Μπορείτε παρακαλώ να μου δώσετε περαιτέρω εξήγηση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κάντενμπαχ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε Σεύκοβιτς, σήμερα είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βασίζεται σε πέντε διαστάσεις και το στρατηγικό πλαίσιο θα καθοριστεί με διάφορα μέτρα. Δεν αναφερθήκατε σήμερα στην πυρηνική ενέργεια σε κάποια από αυτές τις πέντε διαστάσεις. Μεταξύ άλλων κρατών μελών και η Αυστρία απορρίπτουν την πυρηνική ενέργεια και άλλα θέλουν να την καταργήσουν βαθμιαία. Ε, Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσει να υπάρχει η πυρηνική ενέργεια ως σημαντικό μέρος ε, της ε, παροχής ενέργειάς μας. Τίθεται λοιπόν το θέμα της ε, πιο ασφαλούς χρήσης της. Χρειαζόμαστε λοιπόν από τη μία πυρηνική εποπτεία και από την άλλη θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ενεργειακή πολιτική στα κράτη-μέλη. Η σχετική οδηγία ενισχύει τον ρόλο ε, της Κομισιόν στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Ε, μήπως λοιπόν πρέπει να διαχωρίσουμε το ρόλο της πυρηνικής εποπτείας ε, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να μην έχουμε σύγκρουση συμφερόντων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δέμες Μέκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Η πολιτική ενέργεια έχει τρεις αρχές, ότι πρέπει να μπορούμε να την πληρώσουμε, να είναι επίσης αντοχής στο χρόνο και να μην ρηπαίνει. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, εκεί από που έρχομαι εγώ, η Φλάνδρα έχει επιλέξει την γεωθερμική ενέργεια, να τη διευκολύνει. Ένα μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού είναι κατάλληλο για την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας ε, και στο Παρίσι και στο Βερολίνο και σε εμά στην Ολλανδία, στη Φλάνδρα. Εσείς λοιπόν πώς βλέπετε την εκμετάλλευση αυτή σε μεγάλη κλίμακα. Δεν πρέπει να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία να αξιολογηθούν οι οικονομικές συνθήκες και τα ρίσκα. Εσείς από τις αρχές της χρονιάς ξέρετε ότι υπάρχουν ζητήματα με την τιμή της ε, ηλεκτρικής ενέργειας στο Βέλγιο. Δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ στην υπόλοιπη Ευρώπη, εδώ όμως στο Βέλγιο ναι. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τις επενδύσεις. Πρέπει να δούμε λοιπόν και να συντονίσουμε την ε, ζήτηση με την προσφορά και όλο και περισσότερο να προωθούμε την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων και να τα προωθήσουμε. Άκουσα ότι υπάρχουν Νορβηγοί εδώ στην αίθουσα. Λοιπόν, στην Νορβηγή ήταν το όχημα που πουλήθηκε περισσότερο. Είναι μια αμερικανική εταιρεία που βγάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ευχαριστούμε κύριο Σπέτερλε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, με χαρά άκουσα την παρουσίασή σας. Η Ενεργειακή Ένωση είναι απαραίτητη, είναι όμως και ευκαιρία. Δεν τη χρειαζόμαστε μόνο για να αντιμετωπίσουμε ε, αναταράξεις στην, στον ενεργειακό εφοδιασμό, αλλά και για να διαχειριστούμε σωστά τις ενεργειακές πηγές μας. Οι προσπάθειές σας ε, ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε σημαντικές ενεργειακές αρτηρίες Χρειαζόμαστε όμως και μικρότερα αγγεία εντό εισαγωγικών. Χρειαζόμαστε δηλαδή καλό εφοδιασμό και σε τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε μια, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Ακόμα και οι μικροί γεωργοί έχουν λίγο ήλιο, μπορεί να μην έχουν κατοαγελάδες, ο καθένας όμως μπορεί να εκμεταλλευτεί την ηλιακή ενέργεια. Και θα πρέπει να μειώσουμε την ενεργειακή εξάρτηση των γεωργών μας ως μέρος της ενεργειακής πολιτικής μας και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν γι' αυτό και οι σχετικές ενισχύσεις. Τι θα κάνετε λοιπόν κύριε Αντιπρόεδρε για να έχουμε ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό και στην Γεωργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι ενεργειακοί στόχοι για το 2030 είναι καθορισμένοι. Αλλά σε μεγάλο ποσοστό είναι ενδεικτικοί στόχοι. Ο στόχος του 27% της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι κάτι δεσμευτικό για τα κράτη-μέλη. Το ίδιο έχει και το στόχο το γενικό, τον ενεργειακό. Οι στόχοι της Ενδικής Ένωσης έχουν ε, στην ενίσχυση των διασυνδέσεων, βελτίωση της ασφάλειας και να συναφρήσουν τις εθνικές πηγές, όπως είπε και ο Επίτροπος σήμερα. Πώς μπορούμε να πετύχουμε τους ανλόγους στόχους, εάν το ενεργειακό μείγμα ουσιαστικά παραμένει μια επιλογή βασικά εθνική των κρατών μελών. Κάποιες χώρες επιλέγουν την πυρηνική ενέργεια. Άλλες χώρες χρησιμοποιούν τον άνθρακα περισσότερο. Άλλες έχουν πιο πράσινο όραμα όσον αφορά την ενέργεια. Και έχουμε και ιδιαίτερες σχέσεις με τη Ρωσία. Κάποιες χώρες της Ευρώπης προσπαθούν να ενισχύσουν τις σχέσεις με την χώρα. Ξέρουμε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει δρομολογήσει ειδικέ δράσεις γι' αυτό να αυτό. Κάτι που είπαν και συνάδελφοι θα ήθελα να τονίσω κι εγώ. Πιστεύετε ότι όλες αυτές οι διαφορές συνάδουν με την ιδέα μιας ενεργειακής ένωσης. Ποιες συγκεκριμένε δράσεις, όχι μόνο αυτές που αναφέρονται στα έγγραφα, ποιες συγκεκριμένε πράξεις μπορείτε να δρομολογήσετε για να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας για έναν ενεργειακό τομέα ενωμένο στην Ευρώπη. Και κάτι άλλο. Σε ποιο βαθμό και αν θα υποστηρίξετε την έρευνα και τη χρήση των νέων τεχνολογιών για την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σλέκ έχει το λόγο. Uh, uh, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να, να συγχαρώ τον κύριο Σεύκοβιτς για τις προσπάθειές του όσον αφορά τη διαβούλευση όλων των ενδιαφερομένων για να πετύχει όσο γίνεται πιο σύντομα συνένεση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της ενεργειακής κοινότητας το 2005 υπογράψαμε ακριβώς αυτήν την κοινότητα η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από το 2006. Έχει 8 μέλη συνολικά αυτή η Ένωση, τα, τις χώρες της, των Δυτικών Βαλκανίων ε, και την ε, Τουρκία, Νορβηγία ε, ως συνδεδεμένα μέλη. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, θα υπάρξουν τροποποίησεις όσον αφορά τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνυπογράψει αυτήν την κοινότητα και ποια θα είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτήν την κοινότητα, δεδομένου ότι έχουν υπάρξει από διάφορες χώρες προτάσεις για ε, εργοστάσια παραγωγής ρεύματος από άνθρακα, που, κάτι που δεν συμβάλλει στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Πώς μπορούμε λοιπόν να αποτρέψουμε την δημιουργία τέτοιων εργοστασίων Ιδιαίτερα έχοντας υπόψη ότι πολλές από τις χώρες που προτίθενται να δημιουργήσουν τέτοια εργοστάσια είναι υποψήφια προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η ερώτησή μου δηλαδή είναι αυτή. Τι θα κάνουμε με τι εγκαταστάσει ε, παραγωγή ρεύματο από άνθρακα σε σχέση με τον στόχο για την απαλλαγή από θα ακούσει εκπομπέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριο Κόβατσεφ, ε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την παρουσίαση του προγράμματο σα στην Επιτροπή μα σήμερα. Τα τελευταία χρόνια κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επενδύσει πολλά χρήματα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και κάποια κρατημέλη έχουν ξεπεράσει ακόμα και τους στόχους. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές ε, λιανικής της ενέργειας έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η Κομισιόν τι προτίθεται να κάνει για να παραμείνει ελκυστική για τους επενδυτές η πράσινη ενέργεια και τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχει πιο συντονισμένη εφαρμογή νομοθετικών μέτρων στον τομέα αυτών. Και όσον αφορά την μεταβασή ενεργειακών πιστοποιητικών κλπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε για την παρουσίαση σας εδώ σήμερα και που συζητάτε μαζί μας ε, τις ε, προτεραιότητες σας για την Ενεργειακή Ένωση. Και χάρηκα που είδα ότι ε, ένας από τους πέντε πυλώνες της Ενεργειακής Ένωσης στην παρουσίασή σας ήταν ακριβώς η έρευνα και καινοτομία. Διότι ειλικρινά πιστεύω ότι η έρευνα και καινοτομία στον ενεργειακό τομέα θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει περισσότερο την ενέργεια στον τομέα της ενέργειας. Πέρα όμως από το να έχουμε μια τέτοια πρόταση στο χαρτί, σημαντικό είναι να πραγματοποιήσουμε μια τέτοια πρόταση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι δράσεις κλειδιά έχει σκοπό να υποβάλει η Επιτροπή για να εφαρμόσει τον στόχο αυτό όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, τι πλαίσιο έρευνας σκοπεύει να αναπτύξει η Επιτροπή για αυτές τις νέες τεχνολογίες και επίσης θα υπάρξει κάποια ρύθμιση για να ε, έχουμε ομαλή μετάβαση προς μια οικονομία απαλλαγμένη από άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τζάνι, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, και εγώ συμφωνώ με εκείνους που σας ευχαρίστησαν θερμά για την χρησιμότατη συνοπτική παρουσίασή σας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην προσπάθεια οικοδόμησης Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ενώσεως. Αυτή η Ένωση είναι ζωτική σημασία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Αυτό είναι διαμφισβήτητο. Πρέπει να προσφέρει λοιπόν πραγματικά ευρωπαϊκές εναλλακτικέ λύσεις και θα πρέπει να ολοκληρωθεί τάχιστα. κυρίως υπό το φως ανησυχητικών δηλώσεων για τις μελλοντικέ διαθέσεις των Ρώσων. Να θέσω ένα συγκεκριμένο θέμα. Ειλικρινά μιλώντας κύριε Αντιπρόεδρε ανησυχώ τα μάλα όσον αφορά το πόσο υπάρχει πολιτική βούληση σε κάποια κράτη-μέλη να εφαρμόσουν συμπεφωνημένα μέτρα που θα χρησιμεύσουν στην δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης. Υπάρχουν κάποια οράματα στρεβλά σε διάφορα κράτη-μέλη και δεν σέβονται τις βασικές αρχές και υπονομεύουν τις κοινέ προσπάθειες που στόχος είναι εναλλακτικές, ε, βιώσιμες εναλλακτικές πηγές ενέργειας και διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας. Υπάρχει ένα νέο νομοθέτημα στην Ουγγαρία που θεσπίζει πρόσθετη φορολόγηση όσον αφορά τους ηλιακούς ισορρευτές. σε επίπεδο που ίσως ε, δεν προστατεύεται παρακώς και το περιβάλλον, διότι μπορεί να υπάρχει διαρροή από, από ε, μπαταρίες θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε και το PAX 2 που είναι πυρηνικό σταθμό σύμφωνα με αυτή τη λογική, που είναι αντίθετη από τη συμπεφωνημένη στρατηγική. Λοιπόν, προσέξτε κύριε Επίτροπε, χρειάζεται να αποφευθούν τέτοιες πρακτικές πριν να αποδυναμώσουν οριστικά την όλη προσπάθεια. Συνοψίζοντας, εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο μπορούν και πρέπει να συνεργαστούν προς κοινών όφελος. Ευχαριστώ. Κλείνουμε τώρα αυτό το γύρο με τον κύριο Ζουρίνιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήθελα να κλείσω με μία συγκεκριμένη ερώτηση. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την εδώ παρουσία σας. Ανακοινώσατε ότι θα επικεντρώσετε τις προσπάθειές σας επί της υλοποίησης ενός συγκεκριμένου στρατηγικού μοντέλου και βάσει αυτού θα πρέπει να μειωθεί το επίπεδο της αβεβαιότητας. Ένα σημείο που πρέπει να επεξεργαστούμε αφορά τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς. Οι διασυνδέσεις, όπως είπατε, είναι θεμελιώδους σημασία ούτως ώστε να υλοποιηθεί μια αποτελεσματική και ελεύθερη αγορά, αλλά και φυής ενεργειακή αγορά. Το πακέτο για την ενέργεια και το κλίμα, όπως γνωρίζετε, προβλέπει διασυνδέσεις οι οποίες εφαρμόζονται σε δυνητική βάση, δεν είναι υποχρεωτικές. Λοιπόν, Αντιπρόεδρε, πιστεύω ότι στην οδηγία για την Ενεργειακή Ένωση αυτά τα στοιχεία και αυτή η στόχη της διασύνδεσης θα πρέπει να προβλέπονται και να είναι η στόχη υποχρεωτική. Ε, μόνο έτσι θα μπορούμε να έχουμε μια στατική διάσταση που θα είναι ισχυρή και θα στηρίζει το όλο πακέτο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. 23 μέλη έθεσαν ερωτήσεις. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Σεφκοβιτς, για να δώσει απαντήσεις, ευχόμενος του καλή τύχη. Θα τη χρειαστώ κύριε Πρόεδρε, λέει και ο Σεφκοβιτς, αυτό είναι σίγουρο Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις και για τα πολύ καλά σχόλια που κάνατε όσον αφορά τα εισαγωγικά μου σχόλια και τις συστάσεις που ακούστηκαν τι δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε στην τελική μορφή των προτάσεών μας. Θα απαντήσω σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις, ξεκινώντας από την πρώτη ερώτηση της κυρίας Γκροστέτ. Αλλά νομίζω ότι σχετιζόταν εν γέννη με το ερώτημα της κυρίας Μάισνερ και του κύριου Πότς αφορούσε τα δίκτυα, αφορούσε τα ευφυή δίκτυα, τις εθνικές προσεγγίσεις όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική. Όταν σκεφτόμουν ποια θα ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ενεργειακή Ένωση, για να ολοκληρωθεί επιτυχώς αυτή, θεωρούσα ότι η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να αλλάξει η νοοτροπία. Να, η νοοτροπία από εθνική να γίνει ευρωπαϊκή. Συχνά, πολύ συχνά, το αισθάνεσαι αυτό όταν συζητάς τις πολιτικές με τους Υπουργούς Ενέργειας. Βλέπεις πόσοι Υπουργοί Ενέργειας έρχονται στο Συμβούλιο καταρχάς και βλέπεις ποιες σε επικρατούν. Πρέπει να στερνιστούν τη διαδικασία τα κράτη-μέλη. Καλύτερα από πριν. Πρέπει οι Υπουργοί Ενέργειας των κρατών μελών να συμμετάσχουν πολύ περισσότερο, να συμμετάσχουν και οι πολίτες. Πρέπει να ασκηθεί θετική επικοδομητική πίεση που θα οδηγήσει τους Υπουργούς Ενεργείας αλλά και τους Υπουργούς Οικονομίας να κινηθούν. Διότι οι Υπουργοί Οικονομικών είναι πολύ υπεύθυνοι για το τι δαπανάτε για, τις ενεργειακές, για την ενέργεια. Πρέπει να συνεργαστούν, να βρουν ευρωπαϊκές λύσεις. Εδώ μπορείτε να βοηθήσετε εσείς σαν κοινοβούλιο. Και στα κράτη-μέλη μπορείτε να βοηθήσετε. Να παρουσιάσετε την πρόκληση να δείξουμε ότι έχουμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας, αλλά πρέπει να παίξουμε σωστά το παιχνίδι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Τώρα αναφερόμενος στις ευφυείς πόλεις και τα ευφυή δίκτυα. Χωρίς ευφυή δίκτυα δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε ευφυείς πόλεις. Συζητούσαμε επίσης και ποιες ήταν οι εμπειρίες μας των... στις συζητήσεις που έγιναν και στο Ταβός και θυμόμαστε την παρουσίαση που έκανε η ABB, μια επιχείρηση που κινείται στις ενεργειακές υποδομές. Και για στόχους υπερβολής έκανα παράδειγμα. Λέει, αν στο παρόν δίκτυο στην Ευρώπη βάζεις πέντε αυτοκίνητα ηλεκτρικά ε, σε ένα δρόμο, υπάρχει κίνδυνος blackout στον δρόμο. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα δίκτυα αντέχουν. Αντέχουν τη ζήτηση και θα πρέπει οι καταναλωτές να ε, είναι σωστοί καταναλωτές. Θα πρέπει να είναι αμφίδρομη η ροή της ενέργειας. Χρειάζεται ευφυής προσέγγιση και από των καταναλωτών. Άρα χρειαζόμαστε ευφυή δίκτυα. Πώς είναι η ερώτηση. Εδώ ακούμε αντικρουόμενες συμβούλες. Η ΕΝΕΛ 40 εκατομμύρια βάζει ευφυείς μετρητές στην Ιταλία για καλύτερη διαχείριση του δικτύου, για να δίδονται σωστές πληροφορίες στους καταναλωτές. Μετά όμως ακούμε ότι υπάρχουν νέες καλύτερες τεχνολογίες που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν. Άρα πρέπει εμείς οι ίδιοι να βρούμε καλές προτάσεις. Πώς να γίνουν πιο ευφυεί τα δίκτυα ούτω ώστε έτσι οι καταναλωτέ να έχουν μεγαλύτερε δυνατότητε, να μπορούν να χειρίζονται καλύτερα την κατανάλωση ενέργεια των σπιτιών του, να χρησιμοποιούν περισσότερο τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Οπότε εκεί θα παίζει ρόλο σημαντικό και η ζήτηση στον ενεργειακό κύκλο. Θα μπορούμε να έχουμε αμφίδρομη κίνηση της ενέργειας, βελτιστοποίηση των ενεργειακών ροών στα δίκτυά μας, ούτως ώστε να συνεχίσουμε με ηλεκτροδότηση των μεταφορών, ηλεκτροδότηση των αυτοκινητοδρόμων και ούτω καθεξής. Μεγάλο έργο, βασικό, να βρούμε τη σωστή απάντηση. Αν αναφερόμαστε στις ευφυείς πόλεις, τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Πρώτα απ' όλα, ευφυή κατανάλωση ενεργείας. Μετά, ευφυείς μεταφορές. Θα χρησιμοποιεί κανείς δημόσιες μεταφορές, κυρίως αυτές που δεν εκπέμπουν διοξίδιο του άνθρακα, πιθανότατα ηλεκτρικές, ηλεκτροκινούμενες μεταφορές. Άρα προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν να αναπτύξει κανείς και να χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες. Σαφώς πρόκειται περί προκλήσεως προς αντιμετώπιση. Πρέπει να γίνουν πιο ευφύη τα δίκτυα. Κάποιοι από εσά, αρκετοί από εσά, έθεσαν το θέμα της ενεργειακής απόδοσης τι μπορούμε να κάνουμε με τα κτίρια και ότι 80% των κτίριων μας ήδη είναι απειρχιωμένο. Ευαίσθητη κατάσταση. Οι δήμαρχοι και οι πόλεις από τη μια θέλουν να κάνουν περισσότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θέλουν να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουν να γίνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ακούγονται και φωνές που ζητούν σύνεση από διάφορες πλευρές της Ευρώπης μας. Λένε, κοιτάξτε, υπάρχει αρχή της επικουρικότητας. Πρέπει αυτά να θεσπίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο και σε δημοτικό επίπεδο. Η άποψή μου είναι ναι. Έτσι πρέπει να γίνει. Είναι σημαντικότατο ζήτημα. Στις πόλεις μας έχουμε 80% Ευρωπαίους που ζουν εκεί. Και όλα τα προβλήματα ε, συμφόρηση, ρήπανση, τα προβλήματα σύγχρονης ζωής, όλα αυτά που αφορούν το περιβάλλον επικεντρώνονται και περιστρέφονται γύρω από τις πόλεις. Αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε αλλαγή, χρειαζόμαστε και τις πόλεις να συμμετέχουν. Και έχουμε 6.000 δημάρχους που θέλουν να συνεργαστούν. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό, να τους πριζώσουμε τους υπήν στη διαδικασία. Το συζήτησα αυτό με τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Να το συζητήσω μάλλον. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώ να βοηθήσουμε για να κινηθούμε ταχύτερα. Μου είπε όταν το συνάντησα ότι έχω καλή εμπειρία με την, τα προγράμματα στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία για την αποδοτική κρίση τη ενέργεια. Θα το διερευνήσουν περαιτέρω. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, χρησιμοποιώντα τη δυνατότητα που προβλέπεται για να ενθαρρύνει τις, τους Δήμους να επιλέξουν πιο φιλόδοξα προγράμματα. Όταν συζητά κανείς με δημάρχους, μεσαίων και μικρών πόλεων, αυτοί τι λένε. Λένε τα κατάφερα πολύ καλά με τα νοσοκομεία μου, με τα σχολεία μου. Κάναμε εξοικονόμηση ενέργειας. Μοιράσαμε Τις οικονομίες. Μισά χρήματα πήγαν σε επενδυτές, τα μισά ήταν στα χέρια μου, διότι δεν έπρεπε να πληρώσω τόσα πολλά για το κόστος της ενέργειας. Αλλά ήταν νοσοκομεία και σχολεία. Δεν ήταν τόσο μεγάλο το πρόγραμμα. Αν ήθελα να έχω ευρύτερο πρόγραμμα, περισσότερα κτίρια, μεγαλύτερα κτίρια, ήδη είναι μεγάλο το εγχείρημα και φοβούμαι να το κάνω αυτό. Διότι χρειάζονται σύμβουλοι, χρειάζεται η σύμβουλη, χρειάζεται κεφαλιακή επένδυση. Άρα εξυπηρετούμε τους πολίτες τις πόλεις και τους δήμους αν μπορέσουμε να προσφέρουμε τις συμβουλές αυτές πώς να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους, να στηρίξουμε μέσω κεφαλαίων ούτω ώστε να υπάρξει η αναγκαία ανάπτυξη και προσέγγιση στην Ευρώπη. Και πιστεύω ότι μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο μέσο που θα ρίνει και θα προωθεί τέτοια προγράμματα για ενεργειακή απόδοση και σχετικά προγράμματα. Ο κ. Παουλούτσι αναφέρθηκε στο σύστημα ETS και έλεγε ότι πρέπει να προσέξουμε τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Αυτό είναι κάτι που αφορά πολλές περιοχές στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι υπέστησαν πολλές εντάσεις και πιέσεις και καταλήξαμε στα μέτρα για τη διαρροή του άνθρακα που προλαμβάνουν τις εταιρείε. Δεν τις αφήνουν τις εταιρείε να θεωρήσουν την παπάνε αλλού στον κόσμο, σε άλλα μέρη για να έχουν καλύτερες συνθήκες. Όχι, τις δημιουργήσαμε ιδιαίτερες ειδικέ συνθήκες για την πρόληψη διαρροής του άνθρακα. Διάφορα μέτρα θεσπίστηκαν γι' αυτό. Και νομίζω ότι υπάρχει πλέον η αντίληψη ότι αυτό θα συνεχιστεί και μετά το 2020. Το σημαντικότερο, που είναι και συμπληρωματικό, άλλο ένα επιχείρημα, γιατί χρειαζόμαστε συμφωνία στο Παρίσι. Αν πετύχουμε μια γενική συμφωνία, για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, μειώνοντας εκπομπές του διεξουδίου άνθρακος, αυτό σημαίνει ότι θα επικρατήσουν τελικά και ισότιμες συνθήκες για τις επιχειρηματίες μας στο παγκόσμιο προσκήνιο. Η Ευρώπη δεν θα είναι μοναχικός ηγέτης στην πολύ αξιέπαινη αυτή προσπάθεια. Θα συμμετάσχουν και οι ανταγωνιστές μας και οι εταίροι στον κόσμο στη σημαντικότητα αυτή προσπάθεια. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να πετύχουμε καλούς φιλόδοξους στόχους και αποτελέσματα στο Παρίσι. Είναι καλό για τον πλανήτη και καλό για την εξίσωση των συνθήκων που επικρατούν για τους επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο σε διασυνοριακό επίπεδο. Ετέθησαν διάφορα θέματα που αφορούσαν σημαντικότατα προγράμματα για τον ασφαλή εφοδιασμό σε ενέργεια όπως τη Βόρεια Θάλασσα, τη Μεσόγειο και εδώ εξετάζουμε το πώς μπορούμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία που έχουν αυτές οι πηγές ενέργειας. Είναι σαφέστατο ότι βλέποντας την παρούσα κατάσταση και τις σχέσεις με τη Ρωσία και την Gazprom διαπιστώνουμε τη μεγάλη σημασία της ποικιλομορφία της ενεργειακής. Χρειάζεται μεγαλύτερη επιλογή όσον αφορά τις τιμές και την προέλευση της ενέργειας. Ο κ. Μπάκου με ρώτησε την επίσκεψη στη Μόσχα. Ήταν ανοιχτή και ειλικρινή η συζήτηση που έγινε σε όλα τα επίπεδα. Από πολιτική πλευρά αισθανόταν κανείς ότι υπάρχει ανάγκη και επιθυμία για επανέναρξη του διαλόγου για την ενέργεια. Από την άλλη πλευρά του έλεγα σαφώς ότι θα μας άρεσε να το κάνουμε αυτό. Φτάνει να βλέπαμε απτή πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή συμφωνίας του Μίνσκ. Αν βλέπαμε ότι η κλιμάκωση των εντάσεων θα σταματήσει, ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για τη σταδιακή εξομάλυνση των σχέσεων Ουκρανίας-Ρωσίας και Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δυστυχώς βλέπετε τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες Συμβαίνουν πράγματα που δυσχεραίνουν εξαιρετικά την κατάσταση. Ταυτόχρονα η ανακοίνωση του Προέδρου της Gazprom ήταν κάτι άλλο που προξένησε μεγάλη έκπληξη και επιβεβαίωσε ότι υπάρχει κάποια μετακίνηση σχετικά με το σχεδιασμό της Gazprom και πώς επικοινωνεί η Gazprom με τους πελάτες. Δεν μιλάει μαζί τους άμεσα, αλλά μέσω συνεντεύξεων τύπου μετά την αρχική ανάλυση των προταθέντων, δηλαδή 63 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα που περνούσαν από την Ουκρανία από κεντρική δυτική Ευρώπη, αυτά θα διχετευτούν, αυτές οι ποσότητες θα περάσουν από την Τουρκία. Αυτό δεν θα λειτουργούσε σαν πρόταση, δεν είναι οικονομικά βιώσιμη λύση, δεν υπάρχει τέτοια ζήτηση για τέτοιο όγκο αερίου σε αυτή την περιοχή. Η Τουρκία θα χρειαζόταν άλλα 15 BCM δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, άρα, άρα 13 Ευρώπη, 30. Τα άλλα 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα τι θα κάνουμε. Αν μας πούνε κάποιοι θα τα πάρουμε από τον, από τον αγωγό, από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, είναι κάτι διαφορετικό. Η παράδοση γίνεται συγκεκριμένα μέρη και δεν είναι στα ελληνοτουρκικά σύνορα που περνάει ο αγωγός. Ήταν πολύ ισχυρή η δήλωση αυτή, αλλά ελπίζω ότι θα επιστρέψουμε στη συζήτηση για να βρούμε κάτι που θα είναι οικονομικά βιώσιμο, και ρεαλιστικό εντωμεταξύ. Πρέπει να σας πω ότι πρέπει να εργαστούμε ώστε να χρησιμοποιούμε πολλές μορφές ενέργειας, προσπαθούμε να βρούμε νέες πηγές ενέργειας, εφοδιασμού ε, σε φυσικό αέριο από τον νότιο διάδρομο. Θα έχουμε σημαντικότατη συνάντηση στο Βακού όπου θα συναντηθούμε με τον Όμιλο, με το Consortium και θα δούμε ποια θα πρέπει να είναι τα προγράμματά μας, ποιο θα είναι το σχέδιο δράσης, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι ο αγωγός θα κατασκευαστεί έγκαιρα και θα φέρει νέο φυσικό αέριο από νέα πηγή προς την Ευρώπη και τι μπορούμε να διασυνδέσουμε το ευρωπαϊκό σύστημα φυσικού αερίου με τον αγωγό αυτό για να έχουμε περισσότερες επιλογές. Το ίδιο ισχύει και με το φυσικό αέριο, την πλατφόρμα για τη Μεσόγειο υπάρχουν νέες δυνατότητες ώστε το φυσικό αέριο να έρχεται σε μεγαλύτερες ποσότητες από την Αλγερία. Έχουμε νέες πηγές στην Κύπρο, διερευνούμε δυνατότητες για αέριο από το Ισραήλ. Υπάρχουν νέες δυνατότητες να εφοδιαστεί η Ευρώπη σε φυσικό αέριο. Χρειαζόμαστε ενιαία θέση, μία φωνή στη διπλωματία μας, πάρα πολύ ευελικτή υποδομή για το φυσικό αέριο, ποικιλομορφία πηγών και να βελτιωθεί η ελεύθερη ροή του φυσικού αερίου μεταξύ κρατών μελών. Πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη. Εάν χρειαστεί, αν υπάρχει δυσκολία για κάποια κράτη-μέλη, σαν ένωση έτσι θα είμαστε πολύ ισχυρότεροι από ό,τι πριν. Μετά, ο κύριος Κλοντ Τούρμες έθεσε ένα άλλο ερώτημα. Αυτό αφορούσε το νομοθετικό μας πρόγραμμα. Γνωρίζετε ότι ήμουν υπεύθυνο για διοργανικές σχέσεις κατά το παρελθόν, οπότε ξέρω πώς λειτουργεί η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πόσο σημαντική είναι. Συνοψίζω συντομότατα, διότι σύντομα θα συζητήσουμε όταν θα σας δώσουμε τον οδικό χάρτη. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την νομοθεσία για την οδηγία για τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας, για την αποδοτική ενέργεια, ε, οικολογική σήμανση και τα κτίρια και θα πρέπει να προτείνουμε και στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τη θέρμανση και αυτό που ανέφερα. Το μέσο εφιούς χρησιμοποιήσεως για ευφυή κτίρια. Αυτό είναι μια πρώτη γεύση αυτών που θα θέλαμε να προτείνουμε. Αναμένουμε βέβαια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει όπως του αρμόζει, ότι τακτικά θα συμμετέχει στην συνομοθετική διαδικασία και θα βασιζόμαστε όχι μόνο στο να παίξει τον πλήρη ρόλο του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτές τις πολύ σημαντικές προτάσεις. Να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε όσον αφορά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ενώσεως. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ και σε άλλα θέματα που εφήγησαν. Αφορούσαν τις διασυνδέσεις. Βλέπετε ήδη, θα δείτε κάποια πρώτα αποτελέσματα τέλος Φεβρουαρίου που θα εκδώσουμε την πρώτη ανακοίνωση. Πώς θα πετύχουμε δηλαδή 10% διασυνδέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι το 2030 έχουμε πιο φιλόδοξους στόχους και θα πρέπει να καταβάλουμε τις κατάλληλες προσπάθειες. Σημαντικότατο θα ήταν να χειριστούμε καλύτερα ε, τους αγωγούς του προγράμματος. Ήδη το ανέφερα στον πρώτο γύρο των απαντήσεων. Θέλουμε σαφέστατη εικόνα. Τι σχεδιάζεται για ποια χώρα. Ποια πρόοδος έχει επιτεθεί. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, ούτω ώστε να προχωρήσουν τα πράγματα. Τι είναι προβληματικό, τι δεν είναι. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν επικρατεί μόνο η εθνική οπτική γωνία στις συζητήσεις, αλλά εμπεριέχονται και διασυνοριακά στοιχεία διαπιστώνεται και γίνεται αντιληπτή η διασυνοριακή σημασία των προγραμμάτων. Τι ούτω τρόπος θα ξεπεράσουμε τεχνικά και διοικητικά προβλήματα. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Μετά κάποιο άλλο θέμα ετέθη, νομίζω. Ένα ερώτημα που αφορούσε την πυρηνική ενέργεια από την κυρία Κάλενμπαχ. Σαν θεματοφύλακα των συνθήκων πρέπει να σεβόμαστε τις συνθήκες και το σχετικό άρθρο που αφορά την επιλογή των κρατών μελών όσον αφορά το ενεργειακό τους μείγμα. Θα γνωρίζετε βέβαια ότι καταβάλαμε σκληρές προσπάθειες βελτιώνοντας το νομικό πλαίσιο για τον τομέα όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια, διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, προστασία από τη ραδιενέργεια και τώρα θα εξετάσουμε και τα διάφορα επενδυτικά σχέδια για νέους πυρηνικούς σταθμούς και πρέπει οι πυρηνικοί σταθμοί να σέβονται τις πιο τις νεότερες προϋποθέσεις ασφαλείας που έχουν επεξεργαστεί οι εμπειρογνώμονές μας για τα πυρηνικά μετά το ατύχημα της Φούκουσιμα, ούτως ώστε άμα ξανασυμβεί ένα ατύχημα να προστατεύονται οι πολίτες. Ο κ. Τζάνι αναφέρθηκε και στα πυρηνικά καύσιμα και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη διαφοροποίηση των πηγών. Να μην έχουμε προβλήματα τεχνολογικά. Στη Φιλανδία, στο φιλανδικό πρόγραμμα, έργο, ακόμα και αν έχεις ρωσικό αντιδραστήρα μπορείς να έχεις τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές και να βρεις πυρηνικό κάψιμο και από άλλους προμηθευτές. Αν αναφέρεστε λοιπόν σε ποικιλομορφία ενεργειακή όσον αφορά τον εφοδιασμό πρέπει να είμαστε συνεπείς. Να ισχύει η πολυμορφία σε όλες τις πηγές τις ενεργειακές. Και τέλος η ενεργειακή κοινότητα συνεργαζόμαστε πολύ κολλά με το Γενικό Γραμματέα της κοινότητας αυτής. Ήδη αναφέρθηκα στην Ενεργειακή Ένωση. Θα είναι μια ένωση που δεν σταματά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διότι οι γείτονές μας για τις χώρες της ενεργειακής κοινότητας και αυτοί συμμετέχουν στην προσπάθεια, προσβλέπουν στην συνεργασία μαζί μας και προσβλέπουμε και εμείς στην προμόθηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στις εσωτερικές τους αγορές, γιατί έτσι βελτιώνεται η ποιότητα των αγορών τους. Και θα έλεγα ότι βελτιώνεται και η δυνατότητα για καλύτερη ολοκλήρωση των ενεργειακών συστημάτων τους στο ευρωπαϊκό. Σημαντικότατο αυτό που θα είναι τεράστια πρόκληση αλλά σημαντικότατο καθήκον για την Ουκρανία και είναι κάτι που θα βοηθήσει και την Ουκρανία να περάσει αυτή την δυσχερέστατη μετάβαση από πλήρη εξάρτηση από τη Ρωσία μέσω εξυγχρονισμού του ενεργειακού του συστήματος σε πιο ε, αποτελεσματική ε, χρήση ενέργειας με μειωμένη εκπομπή διοξιδίου του άνθρακο, Σε μια οικονομία που θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα να καλύψω τα περισσότερα ερωτήματα που εδέχθην Πιθανότατα να μην απάντησα σε όλους, αλλά ξέρω ότι έχουμε καθυστερήσει λίγο και βλέπω ότι και η Γενική Γραμματεία κοιτάει το ρολόι που μου δείχνει ότι μάλλον πρέπει να σταματήσω εδώ στις απαντήσεις μου. Ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να απαντήσω σε όσου τυχόν δεν σας απάντησα μέσω μικροφόνου. Προσωπικά να σας απαντήσω μπορώ και προσβλέπω και σε μελλοντικέ συζητήσεις μας. Και ελπίζω να έχουμε και την ίδια συζήτηση όταν θα υιοθετηθεί το πακέτο για την Ενεργειακή Ένωση. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε για την παρουσία σας εδώ και σας ξαναπεριμένουμε γρήγορα. Άλλες φορές περιμέναμε για πολύ καιρό. Σας Ευχαριστούμε λοιπόν που σήμερα απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Ταματάμε για ένα λεπτό τη συνεδρίαση προκειμένου να χαιρετήσω τον Αντιπρόεδρο και μετά θα περάσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ. Colleagues, Καθίστε παρακαλώ για να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Okay, so... Uh... Καλώς. Επόμενο θέμα είναι η συζήτηση για μια νέα δασική στρατηγική για τα δάση και το δασικό τομέα. Θα δώσω το λόγο στον ε, συντάκτη γνωμοδότησης, τον κύριο Καμπού. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που μπορώ να σας παρουσιάσω εδώ το σχέδιο γνωμοδότησης όσον αφορά την νέα δασική στρατηγική για τα δάση και το δασικό τομέα. Ελπίζω με τις πολιτικές ομάδες, με τη συζήτηση που θα κάνουμε, να πλουτίσω ακόμα περισσότερο τη γνωμοδότηση αυτή και να ετοιμάσουμε έτσι τη γνωμοδότησή μας για την Επιτροπή Γεωργίας όσον αφορά τα ευρωπαϊκά δάση. Πριν πω στην ουσία θέλω να υπογραμμίσω κάποια σημεία που ίσως να μην τα βλέπετε στη γνωμοδότηση, αλλά είναι ζωτική σημασία. Σήμερα έχουμε 3,5 εκατομμύρια άτομα που απασχολούνται στον τομέα αυτό και 70% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την προστασία της φύσης, που και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να εξακολουθεί να είναι σημαντικό, αλλά έχουμε να κάνουμε και με την συμμετοχή του κόσμου που απασχολείται σε αυτό το τομέα για να βγούμε από την κρίση. Δεν υπάρχει βέβαια κοινοτική αρμοδιότητα, πρόκειται για την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, όχι μόνο σε επίπεδο χωρών, αλλά και σε επίπεδο τοπικό και περιφερειακό, γιατί και αυτές οι αρχές παίζουν ρόλο. Πάντα πρέπει να ξεκινάμε από το πιο κοντινό σημείο στα δάση, να ξεκινάμε από αυτές τις αρχές που βρίσκονται πιο κοντά στα δάση. Προσπαθήσαμε να πετύχουμε ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος, στον κοινωνικό τομέα και τον οικονομικό. Και όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις. Έτσι λοιπόν, επικεντρώσαμε την προσοχή μας στην αηφόρο ανάπτυξη των δασών, ξεκινώντας από μια αρχή αρκετά συνηθισμένη πιο πολύ στα δάση του νότου παρά του βορρά. Και την υπενθυμίζω. Ένα δάσος που δεν καίγεται το καλοκαίρι, προστατεύει καλύτερα από τις βροχές και τις πλημμύρες ε, τον χειμώνα από ότι ένα δάσος που έχει καεί. Γι' αυτό λοιπόν στο πρώτο μου κείμενο θέλησα να συμπεριλάβω την ανάπτυξη ειδικών μέτρων όπως την εισαγωγή της βόσκησης ή τα αγροδασικά μοσαϊκά ως πολιτικές που πρέπει να συμπεριληφθούν στην κοινή γεωργική πολιτική από τον πρώτο πυλώνα που είναι η βόσκηση ή στον δεύτερο πυλώνα που είναι η αγροτική ανάπτυξη και να βρεθούν κίνητρα, για παράδειγμα η πληρωμή για προσφορά περιβαλλοντικών υπηρεσιών, έτσι ώστε και ο ιδιωτικό τομέα να δραστηριοποιηθεί, γιατί αλλιώ δεν θα το κάνει. Είναι αναγκαίο επίσης, αναπτύσσοντας ε, τα διάφορα προγράμματα διαχείρισης των δασών, τα κράτη-μέλη να μην προσθέσουν γραφειοκρατίε στους ιδιοκτήτες δασών, αντίθετα να τους δώσουν κίνητρα για τη διαχείριση αυτή και να μην εγκαταλείπονται και μένα προστάτευτα τα δάση. Θέλω να επεκταθώ επίσης και στην επεξήγηση της τελευταίας παραγράφου στην παράγραφό μου που λέω ότι αυτός που κάνει τη διαχείριση πρέπει να παρουσιάζει ένα σχέδιο διαχείρισης. Έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας τις εμπειρίες που έχει η δίκηση αλλά να τη χρησιμοποιήσει αυτή τη δίκηση αυτός ο οποίος διαχειρίζεται το δάσος είναι αυτή η δήλωση ανάληψης ευθύνης. Θέλουμε επίσης να υποφεληθούμε από την ευκαιρία που μας προσφέρει η βιοοικονομία για να φροντίσουμε για μια εφόρα ανάπτυξη, για δάση πράσινης εργασίας και ανάπτυξη των δασών με μια διαχείριση που να βασίζεται στην εγκύτητα και στην ποιότητα. Τα δάση είναι μια ευκαιρία για την προστασία μεγάλου περιβαλλοντικού πλούτου, της κλωρίδας και της πανίδας μας και είναι και πλούτος για την ανάπτυξη της υπαίθρου προκειμένου να μην εγκαταλειφθούν ε, οι περιοχές αυτές και προκειμένου να υπάρξει νέα επιχειρηματικότητα για την διατήρηση και προστασία των δασών μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και περιμένω τώρα τις απόψεις των άλλων πολιτικών ομάδων για να ολοκληρώσουμε μια ισορροπημένη γνωμοδότηση που να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες του σώματος και να αποτελεί μια προσθεθέμενη αξία στην έκθεση επί της ουσίας της κυρίας Κέστιγκερ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή. Παίρναμε τώρα στους σκιώδεις εισηγητές. Ο κύριος Μπρένα έχει πρώτα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο που παρουσίασε την στρατηγική για τα δάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές τροπολογίες. Υπάρχουν εδώ πολλά που μπορούμε να επικροτήσουμε. Το κυριότερο θέμα εδώ είναι τι θα τονίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσουμε περισσότερο την σημασία των δασών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Καθώς και τη σημασία των δασών ε, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό αναφέρθηκε και το επικροτώ. Αυτή τη στιγμή τα δάση απορροφούν το 10% του διοξιδίου του άνθρακο. Παίζουν λοιπόν πολύ σημαντικό ρόλο. Εάν αυξήσουμε την κάλυψη των δασών από 40% σε 45% η Ιρλανδία σκοπεύει να αυξήσει την κάλυψη από 10% σε 18% μέχρι το 2050. Εάν λοιπόν μπορέσουμε να αυξήσουμε την κάλυψη θα μπορέσουμε να δεσμεύσουμε περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα, κάτι που είναι ε, πολύ σημαντικό. Επίσης, με την καλή διαχείριση των δασών ε, δεσμεύουμε περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα. Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, αλλά από ό,τι φαίνεται ότι όσο πιο πολύ φροντίζουμε τα δάση μας, δηλαδή δημιουργία θέσεων απασχόληση, τόσο περισσότερο ε, διοξιδίου του άνθρακα μπορούμε να δεσμεύσουμε. Και επίση δεσμεύεται από πράγματα που κατασκευάζονται από ξύλο, όπω τα ξύλινα γραφεία που έχουμε εδώ. Θα πρέπει λοιπόν όπου μπορούμε να κατασκευάσουμε πράγματα από ξύλο να το κάνουμε. Στον τομέα της τεχνολογίας εξετάζουμε την χρήση ινών ξύλου σε διάφορα προϊόντα όπου δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό ε, στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα ε, κάποια μέρη αυτοκινήτων. Πέρα όμως από τον ρόλο για τη δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα που μπορούν να παίξουν τα δάση μα και τα ξύλινα προϊόντα, θα ήθελα να τονίσω τη δυνατότητα δημιουργία θέσεων απασχόληση. Υπάρχουν όμω ε, και άλλα ωφέλη, όπω είναι τα ωφέλη για την υγεία όταν περνάει κανεί χρόνο στα δάση, την βελτίωση της ε, ποιότητας ε, του εδάφους, Εάν ε, δηλαδή καλλιεργήσει κανείς προϊόντα κάπου όπου υπήρχαν δάση πριν, βελτιώνεται η ποιότητα των καλλιεργιών αυτών. Και επίσης γνωρίζουμε ότι η φύτευση δέντρων μπορεί να εμποδίσει τις πλημμύρες που αποτελούν αυξανόμενο κίνδυνο ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσουμε τον ρόλο μετριασμού των δασών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ε, καθώς και των προϊόντων από ξύλο, καθώς και τη δημιουργία θέσεων ε, απασχόλησης ε. θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου δεν είναι ο σκύλος, είναι τα δέντρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στόρμαν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή Επικροτούμε τη νέα στρατηγική για τα δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα έχουμε ανάγκη από καλύτερο συντονισμό. Υπάρχει μια σειρά πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η ενεργειακή, η περιβαλλοντική και, και η κλιματική που άπτονται των δασών. 3,5 εκατομμύρια των ανθρώπων ε, της 3,5 ε, εκατομμύρια ε, άνθρωποι απασχολούνται στα δάση, είναι δηλαδή ο τρίτος μεγαλύτερος εργοδότης στα δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε σε στρατηγικές, επικροτούμε τη νέα στρατηγική, ωστόσο θέλουμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε συγκέντρωση αρμοδιοτήτων. η αρμοδιότητα των κρατών μελών στον τομέα αυτών θα πρέπει να γίνει σεβαστή και δεν θέλουμε να έχουμε υποχρεωτικά προγράμματα διαχείρισης των δασών. Δεν θα πρέπει να έχουμε ενιαία κριτήρια σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη συζήτηση αυτή και ιδιαίτερα οι εκπρόσωποι του δασικού τομέα. Όσον αφορά την ενέργεια και την καινοτομία θα πρέπει επίσης να λάβουν προτεραιότητα, διότι ο τομέας των δασών μπορεί να υποφεληθεί από νέες ιδέες. Η αυξημένη αστικοποίηση οδηγεί σε διάβρος των δασών και γι' αυτό θα πρέπει να ε, θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία το θέμα των ε, δασών και μια ισχυρή δασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που να προσελκύει την καινοτομία και τις επενδύσεις θα οδηγήσει σε επιτυχία στην μελλοντική βιοοικονομία. Τα σχέδια διαχείρισης των δασών είναι στρατηγικά μέσα για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές δασών και στόχο έχουν την διασφάλιση βιώσιμων δασών με βάση τις εθνικές νομοθεσίες. Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν εθελοντικά εργαλεία για τους ιδιοκτήτες δασών. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Now, uh, Mrs. Ευχαριστώ η κυρία Γιατνιμάκη. Μάκη. Kiitoksia. Haluan Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά του και για το εξαιρετικό σχέδιο που έχει υποβάλει. Γνωρίζουμε ότι η διαχείριση των δασών και τα δάση οδηγούν σε πολλές σκέψεις και γίνουν πολλά συναισθήματα. Υπάρχουν κάποιοι που φοβούνται λίγο τα δάση, κάποιοι που βγάζουν το βιό τους από τα δάση, άλλοι που γνωρίζουν λίγα πράγματα για τα δάση. Όπως ακριβώς ε, ανέφερε ο συντάκτης της νομοδότησης, ε, θα πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας. Ε, θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να υπάρξει κάποιο είδους συντονισμός στις χώρες της Βαλτικής μάλλον στην Μεσόγεια είχαμε πολλές πυρκαγιές στα δάση. Όπως και σε άλλα μέρη είχαμε καταστροφές δασών άλλων ειδών. Μπορεί κάλλιστα ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου να μην είναι ο σκύλος, να είναι τα δάση, να είναι τα δέντρα. Άλλωστε είναι εξαιρετικό υλικό ε, οικοδομών και υπάρχουν πολλές χρήσεις για τα δέντρα. Σε δύσκολους οικονομικά καιρούς θα πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε ότι συνεχίζουν να φυτρώνουν τα δέντρα ακόμα και σε δύσκολες οικονομικά περιόδους. Είναι λοιπόν μεγάλος εργοδότης ε, στην Ευρώπη τα δάση και μπορεί η στρατηγική προστασία των δασών να παίξει σημαντικό ρόλο. Σε πολλές κοινωνίες ε, δημιουργούνται θέσεις εργασίας λόγω των δασών ε, και γι' αυτό έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντική ευθύνη όσον αφορά τα δάση. Είναι πολύ σημαντικά θέματα η βιοπικιλότητα και η διάβρωση των δασών. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που είναι η διατήρηση των δασών και η εκμετάλλευση των δασών. Αυτά δεν είναι απαραίτητα αντιφατικά μεταξύ τους, μπορούν να συνδυαστούν. Εάν λοιπόν έχουμε σωστή διαχείριση των δασών, προστατεύουμε το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό θέμα η ε, στρατηγική προστασία των δασών και είναι πολύ σημαντικό να διαμορφωθεί σωστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κίλονεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Γκάμπους για την ε, ισορροπημένη γνωμοδότησή του. Είμαι Φινλανδή Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε δασική περιοχή. Έχω λοιπόν ισχυρούς δεσμούς με τα δάση μας ε, και πολύ σεβασμό για το θέμα αυτό. Η ξυλία δεν είναι απλά πρώτη ύλη, τα δάση είναι απαραίτητα και για την ευημερία των ανθρώπων και των ζώων και είναι σημαντικά και για την διασφάλιση της βιοποικιλότητας. Κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά ε, είναι σημαντικά τα δάση. Γι' αυτό θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πρώτες ύλε από τα δάση δεν είναι μόνο η ξυλία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το ευρύτερο φάσμα. Τα δάση οδηγούν σε νέες λύσεις, σε περιβαλλοντικά βιώσιμες μας παρέχουν κατοικίες, ε, καύσιμα και άλλα. Πιστεύω ότι η στρατηγική για τα δάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καταφέρνει να βρει την ισορροπία ανάμεσα στις ε, διάφορες διαστάσεις του θέματος. Πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιες βασικές αρχές. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αφήσουμε τις ε, επιμέρους αποφάσεις στο τοπικό επίπεδο αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει δηλαδή να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Επίσης θα πρέπει να έχουμε βιώσιμη διαχείριση των δασών και ανανέωση των δασών. Θα πρέπει να έχουμε σαφείς αρχές για την εφαρμογή όλων αυτών. Και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε σχέση με το περιβάλλον μας. Ελπίζω στο μέλλον, στα διεθνή φόρουμ και στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής να λαμβάνονται υπόψη οι προκλήσεις μιας βιώσιμης διαχείρισης των δασών και σε άλλα μέρη του κόσμου. Είναι σημαντικό για τη διατήρηση της βιοπικιλότητας σε όλο τον κόσμο, καθώς και για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Να θυμόμαστε όταν συζητάμε την ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση, φέρουμε και αυτήν για τα δάση όλο του κόσμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μαξουρώνης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η δασοκομεία και το τομέας της ε, υλοτομίας είναι πάρα πολύ ευάλωτοι τομείς που μπορούν να επηρεαστούν πολύ εύκολα από πολιτικές αλλαγές. Άρα χρειάζεται ένας καλύτερος συντονισμός των δράσεών μας και χρειάζεται συνοχή αυτών. Χρειάζεται και συντονισμός δράσεων με πολιτικές. Η νέα στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει όλη την αλυσίδα του δασοκομικού τομέα μέχρι την διάθεση στην αγορά των διαφόρων σχετικών προϊόντων. Αυτό θα πρέπει να είναι η βασική αρχή. Ορθολογική χρήση των δασοκομικών πόρων θα πρέπει να οδηγήσει σε καλύτερο έλεγχο των περιοχών της υλοτομίας και θα πρέπει να εφαρμόζονται τα δέοντα μέτρα. Αν θέλετε να εφαρμόσετε σωστά τη στρατηγική, χρειαζόμαστε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσεως εστιαζόμενο επί ισόρροπης χρήσεως όλων των πτυχών, ούτω ώστε να δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Ένα μέτρο θα πρέπει να θεσπιστεί προς στήριξη των ιδιωτών ιδιοκτητών δασών και να δημιουργείται ασφάλεια δικαίου για την εφαρμογή την ομοιόμορφη αρχών σχετικών με τη διαχείριση των δασών. Οι ιδιωτικοί εταίροι ούτω τρόπος θα μπορούν να συμμετέχουν στη διαχείριση των δασών σε μια ισότιμη βάση. Ένας άλλος στόχος να εξασφαλίσουμε την, τα μεγαλύτερα οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη από τη σωστή εφαρμογή των μέτρων. Ολοκληρώσαμε, λέει ο Πρόεδρος, με τους κοιόδης ηγητές. Μπορούμε να πάμε στα μέλη. Η κυρία Γκαρθία Πέρεθ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνο με πολλές από τις σκέψεις που ακούσαμε εδώ από τους υπόλοιπους. Το καταλαβαίνω. Σήμερα δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια κοινή πολιτική για τα δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίποτα όμως δεν εμποδίζει τις πλούσιες σε δάση χώρες να είναι αλληλέγγυες με εκείνες οι οποίες χρειάζονται βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσουν τα δάση τους που απειλούνται από τις κλιματικές αλλαγές, τις πυρκαγιές, την ξηρασία. Γι' αυτό και πολύ θετικά αντιμετωπίζουμε την νέα αυτή στρατηγική και ελπίζουμε να ερμηνευτεί σε συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δασών μας. Στα περιθώρια βέβαια που μας προσφέρει η επικουρικότητα, στην οποία αναφέρθηκαν αρκετοί συνάδελφοι. Αυτό που δεν μπορούμε να στηρίξουμε είναι να καταργηθούν τα σχέδια διαχείρισης ανάληψης ευθύνης η φύση, η εγκατάλειψη των γιών είναι κάτι πολύ αρνητικό. Τα δάση τα οποία δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν και εγκαταλείπονται είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να ξεσπάσουν ε, και μάστιγες, αρρώστιες δηλαδή, αλλά και πυρκαγιές. Πρέπει να ξέρουμε ότι και θέσεις απασχόλησης προσφέρουν τα δάση και μας βοηθούν να καταπολεμήσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Γι' αυτό χρειάζονται σχέδια διαχείρισης. Ακούσαμε τα επιχειρήματα και της κυρία Κέστιγερ και του κυρίου Κάμπους και τους ευχαριστούμε πολύ, όπως επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ευαισθησία που δείχνει πάντα στο θέμα της προστασίας των δασών μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Εύη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή που ετοίμασε αυτό το στρατηγικό έγγραφο για τα ευρωπαϊκά δάση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επικαιροποιήσουμε κάποιες πτυχές όσον αφορά τη διαχείριση των δασών σαν Επιτροπή. Πιστεύουμε ότι η οικονομική αξιοποίηση των φυσικών πόρων μπορεί να συμβάλλει στην προστασία τους. Αλλά για να συμβεί αυτό απαιτείται σωστή ισορροπία μεταξύ εκμεταλλεύσεως των πηγών και αξιοποίησεως των υπηρεσιών και των φυσικών συστημάτων. Τα δάση θα πρέπει να θεωρηθούν όχι μόνο σαν πηγή εφοδιασμού πρώτων υλών που θα χρησιμοποιηθούν σε διάφορους βιομηχανικούς τομούς, τομείς, συγγνώμη, αλλά πάνω απ' όλα σαν ένα σύνολο, ε, σύνολο αλληλεξάρτησης διαφόρων οργανισμών και είναι απαραίτητα για την απορρέφηση του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, για την στήριξη των εδαφών, ε, διότι βλέπουμε στην Ιταλία ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τις βροχές και τη μη συγκράτηση των εδαφών. Είναι πολύ σημαντικό για τη χλωρίδα και την πανίδα. Άρα χρειάζεται να ε, ε, ωφελείται από τα φαινόμενα που ρυθμίζει το δάσος και ο άνθρωπος. Η εκμετάλλευση των πρώτων υλών από τα δάση θα πρέπει να ειδωθεί σαν παράγον που δημιουργεί αναταραχή και αν ε, προσθεθεί η αλλαγή του κλίματος, η όξινη βροχή, η ξηρασία και η διάδοση των πυρκαγιών και των παρασίτων, βλέπουμε μια σφαιρική εικόνα των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει το δάσος. Η προστασία των ευρωπαϊκών δασών είναι βασικό μέτρο για την πλήρη υλοποίηση και άλλων κοινοτικών προγραμμάτων, όπως είναι τα δίκτυα Natura 2000 και διαστάσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τις δασοκομικές δραστηριότητε. Από την άλλη πλευρά, κάποιες ευρωπαϊκές πολιτικέ, ε, πολιτικές όπως η υποχρέωση χρήσης βιοκαυσίμων επιτάχυνε καταστροφικές διαδικασίες αποδάσωσης σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές, γεωγραφικά περιοχές. Πρέπει να προστατεύουμε τις δασικές πηγές, όχι μόνο σε κοινοτικό επίπεδο, αλλά εκτός των συνόρων μας. Αυτό είναι ηθική υποχρέωση. Να υπενθυμίσω ότι οι πολιτικές ε, προστασίες των δασών δεν θα πρέπει να είναι εμπόδιο την ανάπτυξη. Κυρίως όταν η χρήση των φυσικών πόρων δεν θα πρέπει να, χρησιμοποιούνται οι πηγές ε, αυτές που προέρχονται από τα δάση να μην τις χρησιμοποιούμε με μειοπική προσέγγιση και κοντόφθαλμη και όχι μακροχρόνια. Χρειάζεται μακροχρόνια θεώρηση. Ευχαριστώ κύριο Στόρβαλτς, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, η συζήτηση είναι άκρος ε, ενδιαφέρουσα. Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουμε εντελώ διαφορετικές εμπειρίες όσον αφορά τα δάση Υπάρχει κάποια ιστορία που ακούγεται. Ένας Ολλανδός διπλωμάτης πλησιάζει ένα Φιλανδό διπλωμάτη. Ο Ολλανδός ρωτά το Φιλανδό. Πόσα δάση έχετε στη Φιλανδία εσείς. Δεν την καταλάβαινε κανένας Φιλανδός αυτήν την ερώτηση. Δεν μπορεί να μετρήσει στη Φιλανδία δάση. Εάν κάνω μια βόλτα, βγω από το σπίτι μου. Μπορώ να περπατάω σε δάση για τα επόμενα 200 χιλιόμετρα. Ο Φιλανδός ε, διπλωμάτης πού να απαντήσει στον Ολλανδό διπλωμάτη. Και ο Ολλανδός διπλωμάτης είπε υπερήφανα. Έχουμε 18 δάση εμείς στην Ολλανδία. Καλό για αυτούς αλλά όταν ακούς αυτή την ιστορία βλέπεις ότι υπάρχει, ε, λαμβάνεις υπόψη ότι έχεις και σειρματόπλεγμα γύρω τα 18 δάση και υπάρχει λόγος γι' αυτό, να το λάβει αυτό υπόψη. Όταν εξετάζουμε λοιπόν το θέμα των δασών και τη στρατηγική τη σχετική πρέπει να καταλάβουμε ότι μιλάμε για πολύ διαφορετικά πράγματα. Όταν ο, ο φίλος, η φίλη μας αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία για τα δάση στην Ανατολική Φιλανδία αυτή η εμπειρία είναι πολύ διαφορετική από τη δική μου. Ακόμα και αν ε, έχουμε την ίδια χώρα καταγωγής. Δεν σημαίνει ότι κάθε δάσος πρέπει να τεθεί υπό καθεστώς προστασίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ας αφήσουμε τα δάση εκεί στην ησυχία τους για μας. Ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Η στρατηγική για τα δάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προωθεί μια σφαιρική προσέγγιση και τη μετώπιση των δασών με πολλαπλά ωφέλη ενσωματώνει θέματα εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής δασών και λαμβάνει υπόψη την αξία των δασών. Έχει και μια ισορροπία ανάμεσα στην προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην εθνική ευθύνη ευθυγραμμιζόμενη με την αρχή της επικουρικότητας. Η στρατηγική αναγνωρίζει ότι πέρα από τις παραγωγικές λειτουργίες υπάρχουν ε, και άλλες υπηρεσίες οικοσυστήματος και γενικότερα κοινωνικά ωφέλη από τα δάση. Πράγματα τα οποία ανέφεραν διάφοροι ομιλητές, είτε είναι οικότοποι ζών, είτε είναι προστασία, ε, καθαρό κλίμα, ε, εκπομπές του άνθρακα που εξουδετερώνονται κλπ. κλπ. Είναι λοιπόν ζωτική σημασία στις δασικές δραστηριότητες να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι περιορισμένοι οι πόροι και ότι αν δεν θέλουμε να υποβαθμιστούν πρέπει να τα προστατεύουμε. Συνεπώς έχουμε μια ευκαιρία για μια αηφόρο οικονομία στην Ευρώπη που να βασίζεται στα δάση και τα δασικά προϊόντα. Πρέπει να προσέξουμε το ρόλο των δασών στις κλιματικές αλλαγές και από την άλλη όμως να έχουμε υπόψη μας πόσο ευάλωτες είναι οι κλιματικές αλλαγές ξηρεσία, πυρκαγιές, ασθένειες καταστρέφουν πολύ εύκολα τα δάση. Συνεπώς πρέπει τη παραγωγική λειτουργία των δασών με την προστασία τους να τα συνδέσουμε λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δασών. Περιμένουμε τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσβλέπουμε στη συζήτηση και στο τελικό κείμενο που θα βασίζεται στις επιτροπές ΕΝΒΙ, Ήτρε και ΆΓΡΙ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκαμπούς, τον ε, συντάκτη της γνωμοδότησης για τα συμπεράσματά του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια όλους τους συναδέρφους. Το είπα και στην αρχή ότι ήθελα να πετύχω μια ισορροπία. Γιατί αρχίσαμε τη σύνταξη της νομοδότησης αυτής έχοντας υπόψη ότι πρόκειται για μια πραγματικότητα που διαφέρει από χώρα σε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό φάνηκε και από τις παρεμβάσεις των συναδέρφων. Μπορούμε να μιλήσουμε για συντονισμό, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ομοιογένεια. Ακριβώς γιατί η πραγματικότητα διαφέρει από χώρα σε χώρα. Δεν είναι το ίδιο τα δάση της Φιλανδίας όπως είναι τα μεσογειακά δάση ή τα Ολλανδικά. Η βούληση πάντως του συντάκτη σας είναι να πετύχει ακριβώς αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη τα δάση να βοηθούν για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και συγχρόνως να δημιουργούν απασχόληση, οικονομικά ωφέλη και συγχρόνως θελήσαμε να έχουμε υπόψη μας και αυτό ακριβώς το γεγονός των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των χωρών μας όσον αφορά τα δάση. Ευχαριστώ την κυρία Γκαρθία που αναφέρθηκε στην αλληλεγγύη βορρά-νότου όσον αφορά τα δάση. Είπα πριν ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μειογένεια, μια που δεν υπάρχει στα δάση μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν σχέδια δασικής διαχείρισης. Όχι. Τα σχέδια αυτά δασικής διαχείρισης δεν μας εμποδίζουν να κρατάμε ζωντανά τα δάση που αφού είναι ζωντανά είναι καθαρά και αφού είναι καθαρά δεν καίγονται και αφού δεν καίγονται εξακολουθούν να παράγουν και αφού παράγουν εξακολουθούν να είναι χρήσιμα σε όλους για να πετύχουμε τους στόχους μας. Με τα σχέδια διαχείρισης έχουμε ένα καθαρά διοικητικό μέτρο. Και τα δάση τα οποία δεν γνωρίζουμε σε ποιον ανήκουν, καταλήγουν εγκαταλελειμμένα και άρα καίγονται και δεν εξυπηρετούν την επίτευξη των στόχων μας. Δεν λέμε στην γνωμοδότηση να εξαφανιστούν, καθ' άλλο. Απλώς λέμε να χρησιμοποιηθούν πιο στοχευμένα βάσει του τελικού στόχου. Δηλαδή να παραμένουν καθαρά τα δάση και να μας βοηθούν να καταπολεμάμε την κλιματική αλλαγή και να δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης. Είμαι σίγουρος ότι η συζήτηση αυτή και με τις τροπολογίες που θα υποβληθούν θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το κείμενο. Σας ευχαριστώ λοιπόν εκ των προτέρων και όλη αυτή την καλή συνεργασία που θα έχουμε μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκαμπούς. Ωραία. Το χρονοδιάγραμμα είναι ότι η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών 28 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στην Εύβη στις 24 Φεβρουαρίου. Συνεπώς, εδώ λίγη η συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα είναι 5η 29 Ιανουαρίου. Καλό βράδυ.